beginning. I speak Spanish. Buenas tardes. Χαίρετε. Καλώς ήρθατε. Θέλω να σας πω ότι αυτό το θέμα και το επόμενο θα συζητηθούν από κοινού με την ε, αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία. Ινδία. Θα ακούσουμε μια ενημέρωση σχετικά με την επίσκεψη της αντιπροσωπείας ε, στην Ινδία 15 με 18 Μαρτίου. Είναι πάρα πολύ επίκαιρη η συζήτηση αυτή διότι έχουμε αντιπροσωπεία του Ινδικού Κοινοβουλίου ε, υπό την ηγεσία της Προέδρου της Βουλής και επισκέπτεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι δύο επισκέψεις για να επανακτήσουμε και να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας με τα κοινοβούλια μετά τις εκλογές που έγιναν στην Ινδία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευρά μα θέλουμε να έχουμε ενεργή συνεργασία που να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των λαών μα. Να συνεργαστούμε για να επιδιώξουμε κοινού στόχου και αξίε, ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζουμε παγκόσμιε προκλήσει και ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντο. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δώσω το λόγο στον κύριο Τζέφρι Βανόρντεν που είναι πρόεδρος ε, για την αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία για να μας ενημερώσει ε, για την επίσκεψη της αντιπροσωπείας. Έχετε το πολύ 10 λεπτά. Uh, thank uh, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Έχετε δίκιο. Όντως ε, έχουμε την κυρία Σουμίτρα Μαχατζάν μαζί μας η οποία είναι η πρόεδρος της κάτω βουλής του Ινδικού Κοινοβουλίου της ΛΟΚ Σάμπα και θα συνεδριάσουμε αύριο με την παρουσία της κυρίας Μαχατζάν στα πλαίσια της αντιπροσωπείας για τη σχέση με την Ινδία. Θα ήθελα λοιπόν να την καλωσορίσω, καθώς επίσης και τα υπόλοιπα μέλη της αντιπροσωπείας. Όντως έγινε μία αποστολή στην Ινδία από τις 16 έως 18 Μαρτίου 2015. Ήταν ε, η πρώτη τέτοια επίσκεψη που είχαμε εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα και ακολουθώντας τους κανόνες του Κοινοβουλίου φροντίσαμε να κάνουμε μια σύντομη επίσκεψη και να πάμε λίγοι βουλευτές στην Ινδία. Ήμουν λοιπόν εγώ παρόν, οι δύο αντιπρόεδροι, η κυρία Γκίλ και η κυρία Βαν Νόιχεν Χέιζεν, καθώς επίσης και τρεις ακόμη ευρωβουλευτές από την αντιπροσωπεία, οι οποίοι εκπροσωπούσαν συνολικά τέσσερις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, συνολικά μπορούμε να πούμε ότι ε, η όλη επίσκεψη ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική και θετική για να δούμε λίγο το γενικότερο πλαίσιο της επίσκεψης αυτής. Θα θυμάστε ότι δεν είχε γίνει σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας εδώ και πολλά χρόνια και ότι επίσης η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου καθώς επίσης ε, και η Συμφωνία για τις Επενδύσεις και το Εμπόριο η οποία την οποία αρχίσαμε να διαπραγματευόμαστε πριν από 7 χρόνια, έχει φτάσει σε ένα διέξοδο αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε σημειώσει αρκετή πρόοδο τελευταία όσον αφορά λοιπόν αυτή τη συμφωνία. Όταν προγραμματίζαμε λοιπόν την επίσκεψη αυτή, ελπίζαμε να δώσουμε μια κάποια ζωτικότητα στις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδίας. Και ιδίως ελπίζαμε ότι θα μπορούσε να οδηγήσει η επίσκεψη αυτή σε μια σύνοδο Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Ένωση-Ινδία και ελπίζαμε ότι θα λάμβανε χώρα στις 16 Απριλίου, μετά από ένα μήνα δηλαδή. Πάντως, για να συντομεύω θα πω το ακόλουθο. Επίσημω, ήταν η Ινδία αυτή η οποία ακύρωσαν τη Σύνδο. Το κάνω όμω αυτό γιατί νόμιζαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε δαπανίσει πάρα πολύ χρόνο απαντώντας τους και επιβεβαιώνοντας την ημερομηνία τελικά της Συνόδου. Και δίσταν διαπόψεις όσον αφορά την αιτιολόγηση αυτής της καθυστέρησης και υφίσταται και όλο το ζήτημα με τους Ιταλούς πεζοναύτες, το οποίο επηρέασε την όλη κατάσταση. Ένα διμερές δηλαδή πρόβλημα μεταξύ Ιταλίας και Ινδίας, κλώνησε τις γενικότερες σχέσεις ε, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ινδία. Οφείλω να σας πω βέβαια ότι όταν πήγαμε στην Ινδία δεν είχα την πρόθεση να αναφερθώ στα ζητήματα αυτά διότι γνώριζα ότι ήταν ευαίσθητα. Ήδη όμως από την αρχή των συναντήσεων της αποστολής μας στο Δελχή συναντήσαμε εκπροσώπους του τύπου και από ό,τι φαίνεται οι περισσότεροι δημοσιογράφοι θέλανε να μάθουν για ποιο λόγο ακυρώθηκε η προβλεπόμενη σύνοδος. Και αυτό τελικά απασχόλησε ιδιαίτερα τον τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και αυτό ήταν ιδιαίτερα τυχές θα έλεγα. Ωστόσο, συνεχίσαμε προφανώς την επίσκεψή μας στην Ινδία. Λάβαμε ενημέρωση από διάφορους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δελχή, από την επίσημη αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από πρέσβεις από τα κράτη-μέλη της Ένωσης, οι οποίοι βρίσκονται στο Δελχή. Τους ρώτησα βέβαια αν τους αν ρώτησαν τη δική τους γνώμη όσον αφορά την ακύρωση του συνόδου και, της Συνόδου και μου απάντησαν αρκετά εκνευρισμένο ότι κανείς δεν είχε έρθει σε επαφή μαζί τους. Mm. Μας ενημέρωσαν λοιπόν οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ινδία για τις σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Ινδίας. Αναφέρθηκαν λίγο στον απολογισμό του πρώτου έτους της κυβέρνησης Μόντι, το πώς βελτιώνεται ή μπορεί να βελτιωθεί περισσότερη περιφερειακή συνεργασία στην Ινδία, τις γνώσεις που υφίστανται ή την έλλειψη πολλές φορές ενημέρωσης και γνώσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να βρεθήκαμε επίσης και στη δημογραφική πρόκληση της Ινδίας όπου κάθε χρόνο πρέπει να δημιουργούνται επιπλέον ένα εκατομμύριο θέσεις απασχόλησης. Αυτό το στόχο έχουν θέσει οι πολιτικοί της Ινδίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν τα δικά μας προβλήματα μοιάζουν πολύ μικρά σε σχέση με τις δικές τους προκλήσεις. Πήγαμε, όπως σας είπα, στη Λοκ Σάμπα, στην κάτω βουλή του Κοινοβουλίου. Συναντηθήκαμε με την πρόεδρο της κάτω βουλής και έτσι είχα και τη δυνατότητα να την προσκαλέσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και προφανώς, όπως βλέπετε, ανταποκρίθηκε θετικά και ήρθε. Και όχι μόνο αυτό. Καταλήξαμε και συμφωνία να δημιουργηθεί και στην Λοξάμπα μια ομάδα φιλίας Ινδίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και αυτό είναι ένα θετικό βήμα. Συναντηθήκαμε επίσης με μέλη της μόνιμης Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Σασί Τερό είναι επικεφαλής της Επιτροπής αυτής, ενδεχομένως να τον γνωρίζετε ορισμένοι. Είναι πολύ γνωστός, είναι πρώην αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και είχαμε και μια πολύ θετική ανταλλαγή απόψεων μαζί του. Είχαμε και κάποιες επαφές με υπουργούς της κυβέρνησης, τους οποίους είχα συναντήσει και στο παρελθόν, όταν δηλαδή είχαν έρθει ε, στο Δελχή. Μπορέσαμε λοιπόν να τους ε, δούμε. Ο κύριος Νάιντου ήταν παρόν, ο οποίος ασχολείται με την αστική ανάπτυξη, την ε, στέγαση, την εξάλληψη της φτώχειας στα μεγάλα αστικά κέντρα και με τον κύριο Γκατικάρη επίσης συναντηθήκαμε υπουργό αρμόδιος ε, για τις μεταφορές, την αυπηγική και το καθεξής. Ανταλλάξαμε απόψεις με υπουργούς οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τομείς οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντες για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις επενδύσεις και όσον αφορά την περαιτέρω συνεργασία. Πολλές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρονται για τους τομείς αυτού στην Ινδία. Με τον κύριο Κουμασίν επίσης συναντηθήκαμε, ο Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων, ο οποίος αντιμετώπισε πολύ θετικά τις σχέσεις Ινδίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχαμε μια πολύ επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων μαζί του. Συναντηθήκαμε επίσης με τον αναπληρωτή σύμβουλο για αμυντικά θέματα και συζητήσαμε θέματα περιφερειακής αμυντικής συνεργασίας και αναφέρθηκα και σε μία ειδική ευαισθησία όσον αφορά κάποια μέτρα καταπολέμησης της πειρατείας στη θάλασσα. Και αυτό το οποίο μας είπανε ήταν ότι θεωρούσαν ε, ότι είχε επεκταθεί ιδιαίτερα προς τα ανατολικά, πάρα πολύ προς τα ανατολικά, η περίοδος αυτής επαγρύπνησης ή ύψης του αν θέλετε στην αγερμό όσον αφορά την πειρατεία. Και αυτό είχε προκαλέσει ορισμένες φορές διάφορα προβλήματα στις Ινδικές αρχές. Είχαμε επίσης τη δυνατότητα να ε, επισκεφθούμε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικότητας το οποίο ασχολείται με διάφορες δραστηριότητες, κυρίως για την επεξεργασία των υδάτων, τη διαχείριση της ρήπανσης, τις καθαρές μορφές ενέργειας, με τέτοια δηλαδή ζητήματα και προβλέπεται για τους τομείς αυτούς και μια κοινοτική χρηματοδότηση. Επίσης ε, μας ενημέρωσαν εκ μέρους της ΕΚΟ, της Υπηρεσίας δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανθρωπιστική ε, Βοήθεια, μας ενημέρωσαν λοιπόν για τις δραστηριότητες τους σε ορισμένες περιοχές της Ινδίας. Συζητήσεις επίσης κάναμε και με μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας, ε, κατά τη διάρκεια ενό πολύ καλού γεύματος εργασία, καθώ επίση συζητήσαμε και με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας των Εμπορικών Επιμελητηρίων της Ινδία και με εκπροσώπους σημαντικών Ινδικών επιχειρήσεων και συζητήσαμε μαζί τους για κάποιες δυσκολίες που αντιμετωπίσουν αλλά και για τα επιτεύγματά τους, τις σημαντικότερες επιτυχίες τους. Συναντηθήκαμε όμως και με οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών. Δεν ήταν ιδιαίτερα εκτενής η συνάντηση που είχαμε, μολονότι εκπροσωπήθηκαν πολλές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες μας εξέθεσαν τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν μα είπαν ότι δέχονται πιέσεις και ότι τους έχουν επιβληθεί κάποιοι περιορισμοί στη δραστηριότητά τους. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ορισμένες από τις οργανώσεις αυτές ασχολούνται περισσότερο με ομάδες πολιτικής πίεσης τελικά, εκφράζουν περισσότερο πολιτικές απόψεις και ασκούν πολιτική επιρροή και δεν ασχολούνται τόσο πολύ με την ανθρωπιστική δράση. Πέρα όμως από το Δελχή, από το Νέα Δελχή, είπαμε ότι θα πρέπει να πάμε και σε κάποιο άλλο κρατήδιο, σε ένα κρατήδιο το οποίο θα είχε τουλάχιστον κυβέρνηση από το BJP. Αποφασίσαμε λοιπόν να πάμε στο Τζαϊπούρ της Ρατζαστάν Ξέρω εκεί πέρα τους, τον, επικεφαλής, τον επικεφαλής της ε, περιφέρειας, τον επικεφαλής του κρατηδίου. Συναντηθήκαμε λοιπόν μαζί, καθώς επίσης και με τον επικεφαλής της ε, Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Ρατζαστάν και καταφέραμε κατά αυτόν τον τρόπο να καταλάβουμε λίγο περισσότερο ποιες είναι οι σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ κέντρου και περιφέρειας στην Ινδία. Καταφέραμε να επισκεφθούμε και το νέο, τη νέα μονάδα του JCP στο Τζαϊπούρ. Πρόκειται για μια βρετανική επιχείρηση η οποία έχει σημειώσει πολύ μεγάλες επιτυχίες στην Ινδία και έχουν λοιπόν διάφορες μονάδες παραγωγής στη χώρα. Θελήσαμε πάντως να δούμε πώς καταρτίζουν τους νέους Ινδούς, μάλλον νέες Ινδέες γυναίκες από κάποια πολύ φτωχά χωριά της Ινδίας οι οποίες παρακολουθούν διάφορα προγράμματα κατάρτισης και καταφέρουν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες σε συγκεκριμένους τομείς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε το πρόγραμμα αυτό. Επίσης με το κέντρο εμπορίου περιβάλλοντος είχαμε, με προσώπους του κέντρου αυτού είχαμε επαφές. Πολωνότου λοιπόν ήταν τρίμερη μόνο η παραμονή μας στην Ινδία. Θεωρώ ότι καταφέραμε να έρθουμε σε επαφή με πολλούς διαφορετικούς παράγοντες και εκπροσώπους. Είδαμε ότι όντως υπάρχουν πολύ σημαντικά επιτεύγματα στην Ινδία. Ήρθαμε σε επαφή με την επικεφαλή του Συμβουλίου για να δούμε τελικά τι θα γίνει με τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωση Ινδίας που τελικά θα γίνει ελπίζουμε τον Νοέμβριο του 2015 και όπως σας είπα έχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη την πρόεδρο της ΛΟΚ ΣΑΜΠΑ. Κύριε Πρόεδρο, όπως σας είπα, ήταν πολύ επικοδομητική, θετική και ιδιαίτερα σημαντική η επίσκεψή μας στην Ινδία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την εκτενή σας αυτή παρουσίαση. Θέλω να δώσω το λόγο στην αντιπρόεδρο της αντιπροσωπείας στην αρχή συζήτηση, την κυρία Νίνα Γκίλ. Έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με όλα όσα είπε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας. Ήταν πολύ επίκαιρη αυτή η επίσκεψη. Το μικρόφωνο σας, κυρία Αγγίλ, γιατί μιλάτε πολύ μακριά. Μάλιστα. Τώρα με ακούτε. Θα τα πω από την αρχή έλεγα ότι ήταν πάρα πολύ επίκαιρη αυτή η επίσκεψη και δυστυχώς, όπως είπε και ο Τζέφρι, ε, είχαμε αυτό το πρόβλημα με τη Σύνοδο Κορυφής, δηλαδή φτάσαμε στο Δελχή κάπως, πώς να το πω, σε ατυχή συγκυρία. Ε, χρειάστηκε να κάνουμε πολλές δημόσιες σχέσεις εκεί για να αποκαταστήσουμε ε, την κατάσταση. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας το εξής. Με αυτό το διάλογο και αυτές τις επισκέψεις δεν θα πρέπει να επιδιώκουμε μόνο διακοινοβουλευτικές συνεργασίες, εμείς δηλαδή και η Ινδική Βουλή, αλλά ε, θα πρέπει να τα συνδέουμε και με τις συνόδους κορυφής που είναι και πολλές. Προσβλέπω στη συνεργασία και στην ε, επίσκεψή μας, αλλά και την επίσκεψη ε, της Προέδρου της ΛΟΚ ΣΑΜΠΑ ε, χρειάζεται να γίνει ένας νέος διάλογος και να δοθεί μια νέα όθηση για το πώς διαμορφώνουμε τη σχέση μας με την Ινδία. Είναι πολύ σημαντικό να το προωθήσουμε αυτό. Σήμερα το πρωί ο Μάρτιν Σούλτς είπε ότι προγραμματίζει επίσκεψη του χρόνου, αλλά εγώ έκανα ερώτηση προηγουμένως στην ύπατη εκπρόσωπο, θα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική με την Ινδία για το πώς ε, θα προχωρήσουμε στο μέλλον και τι σχέσεις θα έχουμε και ποια θέματα θέλουμε να προωθήσουμε. Δεν μπορούμε απλώς να επενδύουμε ή να ποντάρουμε στη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου που δεν λέω, είναι και αυτή σημαντική. Αλλά υπάρχει και η γεωπολιτική θέση της ε, Ινδίας και η αναπτυξιακή στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ξέρω ότι το είπε φαντάζομαι και ο πρόεδρος Βαν ε, αλλά θέλω να ευχαριστήσω την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτόπου γιατί κατάφεραν να ε, μας φτιάξουν ένα πρόγραμμα πάρα πολύ καλό. Και χάρηκα που είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε επιτόπου την EBTC ε, που είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας. Ε, πολύ δε περισσότερο που εγώ πρωτοστάτησα στην προσπάθεια πριν από λίγα χρόνια να στηθεί αυτό και θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να το υποστηρίζουμε διότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τις δικές μας επιχειρήσεις, ιδιαίτερα από τα West Midlands που κατάγομαι εγώ, που ε, έχουμε εκεί ε, πανεπιστήμια ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις και προσπαθούν να μπλακούν και να εγκατασταθούν και στην Ινδία. Θέλω να ευχαριστήσω και τη γραμματεία επίσης και τον πρόεδρο Βανόρδεν για την τόσο καλή ε, αυτή η επίσκεψη. Κύριος Χαν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ δεν ήμουν μέλος της αντιπροσωπείας. Ελπίζω να πάω στην επόμενη γιατί φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα. Και χαίρομαι για τις πληροφορίες που άκουσα εδώ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι σημαντική η Ινδία και οι καλές μας σχέσεις μαζί της. Γι' αυτό συμφωνώ με αυτά που είπε η συνάδελφος ότι πρέπει να δοθεί παραπάνω όθηση. Όσο ισχυρότεροι, ισχυρότερες δεσμούς έχουμε τόσο καλύτερο και για μας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις ή παρεμβάσεις. Πάμε στο επόμενο θέμα λοιπόν, που είναι η παρουσίαση της μελέτης με τίτλο «Αξιολόγηση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας και των δυνατοτήτων και την αναγωγόνησή της». Έχω τη χαρά να καλωσορίσω τον ε, συντάκτη της μελέτης, ε, τον κύριο Γκούλσαν Σαστέβα, που είναι πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Διεθνών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Νεχρού της Ινδίας. Όπως είπαμε και το προηγούμενο σημείο είναι πάρα πολύ επίκαιρη αυτή η συζήτηση για τις συστάσεις. Το κοινοβούλιο μας είναι υπέρ των καλών σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας και η Επιτροπή μας θέλει να ζαγωνηθεί η σχέση που ξεκίνησε το 2004. Γι' αυτό ζητήσαμε μελέτη για να δούμε τι λένε εξωτερικοί εμπειρογνώμονες επί του θέματος. Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η μελέτη αυτή και διανεμήθηκε στους βουλευτές. Περιμένουμε να ακούσουμε την παρουσίασή σας, κυρία Σαστέβα. Έχετε αμέσως το λόγο για 10-15 λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές και μέλη της αντιπροσωπείας με την Ινδία. Εξοχότατες, εξοχότατοι κυρίες και κύριοι. It's my privilege to be uh, discussing this. Συζητώντας τη μελέτη αυτή μαζί σας, Χαίρομαι γιατί πριν από μερικούς μήνες μου ζήτησε το Κοινοβούλιο να συντάξω αυτή τη μελέτη και επειδή έχω 10 λεπτά μόνο, ελπίζω μερικοί να την έχετε διαβάσει για να είμαι τηλεγραφικός. Να περιοριστώ δηλαδή μόνο στα κυριότερα. Εξετάζοντας τις σχέσεις της Ινδίας με την Ευρώπη διαπιστώνουμε ότι είναι πολύ παλαιές. Από πριν την επικιακή εποχή και μετά την ανεξαρτησία της Ινδίας. Κατά τον ψυχρό πόλεμο η Ινδία ήταν με τους αδέσμευτους και κοντά στη Σοβιετική τότε Ένωση. Και τότε είχε λιγότερες σχέσεις με την Ευρώπη αλλά συνεχίσαμε να έχουμε διμερείς σχέσεις με χώρες της ε, τώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 90 όμως η αντιμετώπιση της Ινδίας ως προς τον πολυπολιτιστικό και πολυπολικό κόσμο άλλαξε και ταυτόχρονα δημιουργήθηκε μία νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας στην Ασία και θεώρησαν και οι Ευρωπαίοι πολιτικοί ότι σωστό θα ήταν να είχαν περισσότερες σχέσεις με την Ινδία για να είναι πλήρης οι δεσμοί με την Ασία. Βλέπει λοιπόν κανείς ότι άρχισαν να αλλάζουν τα πράγματα από το 90 και μετά. Κοινή πολιτική δήλωση του 1993, διμερείς ε, σχέσεις και λοιπά και σε, ποιες, σε ποιους τομείς, ποιους κάλυπταν αυτές οι συμφωνίες. Πολλά, πολλούς. Πολιτική διάλογη και συνεργασία έχουν τα περισσότερα θέματα συμπεριλαμβάνονται. Λαοί και πολιτισμοί, οικονομική, πολιτική, διάλογο, συνεργασία. Όλα τα σημαντικά θέματα καλύπτονται φαρμακευτικά, ενέργεια, μεταφορές, ε, διάστημα κτλ. Για τα εμπορικά συγκεκριμένα υπάρχουν πολλά θέματα που ενέκριναν και οι δύο πλευρές και μετά προσθέθηκαν κι άλλα. Θέματα ασφαλείας, βιώσιμης ανάπτυξης, έρευνας και αυτό σημαίνει ότι όλες οι πλευρές συμφώνησαν σχεδόν για όλα τα θέματα. Τώρα όμως βλέπουμε ότι από το 2009 συγκεκριμένα η σχέση έχει αρχίσει να χάνει την ορμή της. Ένας λόγος είναι το πάγωμα των διαπραγματεύσεων για τον BTIA, γενική κρίση και η πολιτική παράλυση που σημειώνεται στην Ινδία τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν όμως και νέες ευκαιρίες, διότι και η Ινδία και η Ένωση ανανεώνουν τις ηγεσίε τους. Πάντως η καρδιά των σχέσεων παραμένει η οικονομία. Η Ένωση είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ινδίας και τα τελευταία 15 χρόνια οι επενδύσεις στην Ινδία από την Ένωση είναι υψηλότερες από ό,τι από τις Ηνωμένε Πολιτείε και την Ιαπωνία και την Κίνα συνδυασμένες. Οι μεταφορές τεχνολογίας επίσης είναι κυρίως από την Ένωση και οι διαμεθοριακές επενδύσεις επίσης και η συνεργασία στην έρευνα και την καινοτομία επίσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλο το εμπόριο σε αγαθά και υπηρεσίες αυξάνεται με απόλυτους αριθμούς. Τα ινδικά στοιχεία συγκεκριμένα δείχνουν ότι τα τελευταία 15-20 χρόνια κάθε χρόνο μειώνεται το εμπόριο μεταξύ Ινδίας και Ένωσης. Δηλαδή μειώνεται η σημασία της Ευρώπης για την Ινδία γιατί έχει περισσότερο εμπόριο με την Κίνα και άλλες ασιατικές χώρες. Δεν υπάρχουν, υπάρχουν και νέες ευκαιρίες, ας πούμε γίνονται προτεραιότητα τα θέματα ανάπτυξης και ο, η Ένωση παραμένει σημαντικός μας εταίρος. Η νέα κυβέρνηση έχει ανακοινώσει νέες πρωτοβουλίες, το πρόγραμμα Make in India, Clean India, Digital India, καθαρός γάγκης κλπ και τα κράτη-μέλη της Ένωσης, άρα μπορούν να γίνουν σημαντικοί εταίροι και να συμβάλλουν σε αυτά τα προγράμματα. Αν θέλουμε να δούμε τώρα θέματα άμυνας και ασφάλειας και στρατηγικής συνεργασίας, δεν υπάρχει ακόμα σε αυτά μια καθαρή συνεργασία. Αντίθετα με τη Ρωσία και την ίδια της ΗΠΑ, η Ινδία δεν έχει ακόμη καταλάβει τη σημασία που μπορεί να έχει η σχέση της με την Ένωση σε αυτούς τους τομείς. Και γι' αυτό δεν παίζει σημαντικό ρόλο στην εξωτερική πολιτική της Ινδίας. Οι αυξανόμενες όμως Ινδοαμερικανικές σχέσεις μπορούσαν να ωφελήσουν και την Ένωση. Ειδικά για θέματα άμυνας και ασφάλειας η Ινδία εμπορεύεται, συνεννοείται κατευθείαν με τα κράτη-μέλη και η αγορά των τελευταίων ραφάλ από την Ινδία θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στις σχέσεις αυτές τα προγράμματα των ΗΠΑ, Pivot to Asia και ο μεγαλύτερος ρόλος που παίζει η Κίνα επίσης θα παίξουν ρόλο και θα μπορούσε η Ινδία να γίνει ένα κλειδί, ένα εταίρος κλειδί. Για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας η συνεργασία θα εξαρτηθεί από το πόσο θα παίξει κάποιο ρόλο στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας η Ένωση. Πάντως θα μπορούσε και εδώ να υπάρξει συνένεση, συμφωνία και συνεργασία στα πλαίσια τη διεθνού σύμβαση κατά την καταπολέμηση της Για τους ελέγχου τώρα στις εξαγωγέ. Θα μπορούσαν τα κράτη-μέλη της Ένωσης να στηρίξουν τις προσπάθειες της Ινδίας να γίνει και αυτή η πυρηνική δύναμη αν και δεν είναι εύκολο να υπάρξει συνένεση σε αυτό από την Ένωση αλλά κάποια συνεργασία. Πολλές μεγάλες χώρες μέλη όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ισπανία έχουν υποστηρίξει την Ινδία σε αυτό. Αν μπορεί τώρα η Ινδία να παίξει ένα ρόλο στην κρίση της Ουκρανίας. Δεν έχει άμεση συμφέρον, αλλά ως αποτέλεσμα της κρίσης αυτής η Ρωσία έχει πλησιάσει την Κίνα και αυτό επηρεάζει και την Ινδία. Η θέση του νέου Δελχή υποστηρίζει περίπου τη Ρωσία αλλά παρά τη στρατηγική της εταιρική σχέση με τη Ρωσία θα μπορούσε να παίξει κάποιο ρόλο και για την επίλυση της Ουκρανικής κρίσης, για την παγκόσμια διακυβέρνηση. Αυτό θα είναι μια δοκιμή των σχέσεων Ένωσης και Ινδίας. Αλλά ακόμα υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Εδώ θα μπορούσε να υπάρξει περισσότερος διάλογος για την ενεργειακή ασφάλεια και τις ανανεώσιμες αν και θεωρείται ότι έχουν αντιδιαμετρικά αντίθετες απόψεις η Ινδία και η Ένωση για αυτά τα θέματα, υπάρχει μεγάλη δυνατότητα συνεργασίας γιατί και οι δύο πλευρές προσπαθούν να διαφοροποιήσουν τις πηγές τους και υπάρχει τεράστιος χώρος για συνεργασία στις ανανεώσιμες πηγές ενεργείας. Συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών αναφέρθηκε προηγουμένως. Υπάρχουν δύο εκατομμύρια σύλλογοι εταιρεία ε, κοινωνίας των πολιτών στην Ινδία και συνδέονται πολλές φορές με ευρωπαϊκές οργανώσεις όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην αντιμετώπιση των κλιματολογικών αλλαγών κτλ. αλλά επειδή υπάρχει περισσότερη καχυποψία τελευταία από την Ινδία, οι σχέσεις αυτές Ένωση Ινδίας ως προς αυτές τις οργανώσεις έχουν ενταθεί. Για τη συνεργασία, αναπτυξιακή συνεργασία, η Ινδία εδώ και πολλά χρόνια παίζει ρόλο στην αναπτυξιακή συνεργασία, αλλά τελευταία έχει χορηγήσει περισσότερα κονδύλια για εκπαίδευση από την Αφρική και την υπόλοιπες χώρες της Ασίας. Στο Αφγανιστάν ιδιαίτερα η Ινδία θα παίζει σημαντικό ρόλο, θα είναι παρούσα τουλάχιστον μέχρι το 24-25, δεν έχει προβλέψει ακόμα να τελειώσει την παρουσία της εκεί, στους τομείς της capacity building, εκπαίδευση αστυνομικών, ανώτερη παιδεία, αποκέντρωση και θέματα δημοκρατίας. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επειδή είναι δημοκρατία, η Ινδία είναι ευαίσθητη σε κατηγορίες παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων και εδώ το καλύτερο θα ήταν ο διάλογος. Τώρα μερικά διμερεί θέματα που αφορούν σχέσεις Ινδίας και χωρών Ένωσης. Υπάρχει μια στρατηγική κατανόηση αλλά αυτά λύνονται πάντα διμερώς. Έτσι ας πούμε παραδείγματος χάρη το Ιταλικό ναυτικό παίζει κάποιο ρόλο στην Ινδία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως πολιτικό σώμα που εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες θα μπορούσε να το εξισορροπήσει αυτό μη επιτρέποντας καθαρά διμερεί θέματα να καθορίσουν το πρόγραμμα των σχέσεων Ινδίας Ένωσης. Υπάρχει λοιπόν το θέμα του παγώματος των διαπραγματεύσεων του BTIA που θα πρέπει να ξαναρχίσουν αμέσω και καινούργιοι διάλογοι με, ως προς το Αφγανιστάν, τη θαλάσσια ασφάλεια, τον αναπτυξιακή συνεργασία στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Αλλά γι' αυτό χρειάζονται βέβαια περισσότεροι ανθρώπινοι και χρηματικοί πόροι. Επίσης η Ένωση θα μπορούσε να χορηγήσει το καθεστώς Data Secure Status στην Ινδία μερικές θετικές δηλώσεις για τις προσπάθειες της Ινδίας για τα πυρηνικά έχουν γίνει επίσης από το 12 και μετά και έχουν προγραμματιστεί και άλλες τακτικές συνήθειες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σαντεβά. Θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Βανόρτεν. Ε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή Σαχτέβα για την ενδιαφέρουσα εισαγωγή στη μελέτη. Πρέπει να σας πω ότι δεν είχα καταλάβει ότι συνεχίζεται η μελέτη αυτή είναι ενδιαφέρον αυτό να δούμε και τη δυναμική για το πώς λειτουργούν ε, κάποια πράγματα. Δεν είναι καθόλου κριτική στο πρόσωπό σας, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η μελέτη και με χαρά θα τη διαβάσω. Θέλω να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Ε, στο τέλος τονίσατε την ανάγκη να ε, συνεχιστεί η προσπάθεια για τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών. Εσείς γιατί νομίζετε από ειδική πλευράς ότι υπάρχουν κάποιοι δισταγμοί, ας πούμε, αν υπήρχαν για την FTA, τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου, γιατί και οι δύο πλευρές, πώς να το πω, δεν ξετρελάθηκαν. Ε, ούτε θέλησαν να προωθήσουν έτσι, με ζέση αυτό το θέμα. Ε, πώς το βλέπετε εσείς η Ινδική δισταγμή, για ποιο λόγο. Κάποιος μου είπε όταν ήμουν στην Ινδία ότι είχε επιφυλάξει η Ινδία γιατί είχε κακή εμπειρία στο παρελθόν. Ας πούμε την Νότια Κορέα, εμείς είχαμε μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών, ε, μάλλον και εκείνοι δεν ε, είχαν τα ωφέλη που επιδίωκαν. Και δεύτερον, το μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είδαν ποτέ οι Ινδοί με ενθουσιασμό ως ένα πιθανό μοντέλο ή δυνατό για περιφερειακή συνεργασία στην Νότια Ασία. Δηλαδή το έχουν σκεφτεί ή αν το είχαν σκεφτεί στο παρελθόν το έχουν απεμβολήσει τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Αγγίλ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να αφερθώ στο ζήτημα της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών. Πώς μπορούμε να βγούμε από το διέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Και πιστεύετε ότι υπάρχουν ενδεχομένω τομεί στους οποίους θα μπορούσαμε γρήγορα να καταλήξουμε σε συμφωνία και που θα μας βοηθούσαν για τη συμφωνία αυτή τελικά. Έχετε εντοπίσει τέτοιους τομείς στους οποίους θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Επίσης, μου φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η παρατήρηση που κάνετε για τις σχέσεις με τη Ρωσία. Πού θα τοποθετούσατε εσείς επί του παρόντος τις σχέσεις Ινδίας-Ρωσίας. Επίσης, δεδομένου ότι όσα συμβαίνουν στην ανατολική γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρείτε ότι επηρεάζονται και οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας από την κατάσταση στην Ουκρανία, για παράδειγμα. Θα ήθελα επίσης να δούμε το ζήτημα της παγκόσμιας διακυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδίας. Μας είπατε ότι η Ινδία, αλλά ενδεχομένω και άλλες χώρες, αυτή τη στιγμή καθορίζουν τους παγκόσμιους κανόνες όσον αφορά το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και προφανώς η Ινδία θα συμβάλλει πάρα πολύ και για το EINP και για τις χώρες BRICS και τη μεταξύ του συνεργασία. Δεδομένου το ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα έχουν έντονη συμμετοχή στην Ινδία, πώς πιστεύετε ότι θα διαμορφωθεί η σχέση με τους θεσμούς αυτούς η, ο κύριος Ρέγκορα Ραντζάν, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ινδίας, ενδεχομένως να ενδιαφέρεται για την θέση της Κριστίν Λαγκάρτ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όταν λήξε δηλαδή η θητεία της. Ποια είναι η σχέση λοιπόν της Ινδίας με τους μεγάλους αυτούς οικονομικούς θεσμούς. Ε, βλέπουμε επίσης ότι έχει ενδυναμωθεί περισσότερο η σχέση της Ινδίας με την Ιαπωνία, έχει ενταθεί ο διάλογος με την Κίνα. Πού εντάσσεται στο γενικότερο αυτό πλαίσιο η Ινδία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Χάν. Ευχαριστώ. πολύ καθηγητά για την παρουσίαση αυτή. Ήταν συναρπαστική και πάρα πολύ κατατοπιστική. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα τομέα που ανέφερε και η συνάδελφός μου ε, για το θέμα της Νότιο-Ανατολικής Ασίας, Αφγανιστάν και Κίνα. Τι γίνεται με τις σχέσεις Πακιστάν-Ινδία, υπάρχει καμιά ελπίδα εκεί, κανένα φως. Θέλω να σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση για την ένταξη της Ινδίας στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης. Δεν ξέρω αν το λέτε στην έκθεσή σας. Αυτό θα ήταν θετικό ή αρνητικό ε, στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και αυτή την κρυφή ε, αντιπαράθεση, ας πούμε, συγκαλυμμένη μεταξύ, Ευρωπαϊκή, μεταξύ ΕΠΑ και ε, Εναδειωμένων χωρών. Ο κύριος Τάνοκ, ε, κάτι που είπε ε, ο Τζέφρι Βαν για το ΣΑΡΚ ή ΣΑΦΤΑ. Έχω ακούσει δύο φορές από Ρώσους ότι μετά από τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί της Ρωσίας τώρα βλέπουν μια εναλλακτική λύση διεθνού συνεργασίας ας πούμε ε, ε, για μια τάξη ως λιγότερο δημοκρατικής και πιο αυταρχικής που αναδύεται από την οργάνωση της Σανγκάης αλλά και από την εδραίωση των BRICS. Βέβαια η Ινδία είναι ε, δημοκρατία όπως και η Βραζιλία δεν είναι αυταρχικά καθεστώτα. Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα λοιπόν και άλλοι κάπως συνεργάζονται με τρόπο πιο συνεκτικό, πολιτικό και οικονομικό και με τράπεζα επενδύσεων. Εσείς πώς το αξιολογείτε αυτό, έχει κάποια βάση ή απλώς προσπαθούν οι Ρώσοι να απλοφάρουν και να ε, φοβήσουν τη Δύση για να χαλαρώσουν τις κυρώσεις. Γιατί τι σχέση μπορεί να έχουν όλες αυτές οι χώρες και λιγότερο από όλες η Ινδία και η Κίνα ας πούμε. Αν δεν έχετε άλλες ερωτήσεις παρακαλώ το λόγο έχει ο κύριος καθηγητής για να απαντήσει. Mm. Thank Σας ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες και χρήσιμες ερωτήσεις. Θα τις έβαζα σε δύο-τρεις κατηγορίες τις ερωτήσεις σας. Υπάρχουν ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με το ελεύθερο εμπόριο, άλλες πάλι με τη Ρωσία. Μια ερώτηση έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρότυπο περιφερειακής συνεργασίας για την Ινδία, για τη δική μας δηλαδή περιφέρεια. Θα ξεκινήσω καταρχάς με το τελευταίο αυτό το με Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρότυπος μοντέλο περιφερειακής συνεργασίας. Όντως ανέκαθεν βλέπαμε ως πρότυπο την Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο για την Ινδία και την Ανατολική Ασία αλλά γενικότερα για το στόχο. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που θαυμάζουν την εμπειρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσπαθούν να τη μιμηθούν. Αυτό όμως το οποίο συμβαίνει σήμερα είναι ότι ορισμένοι έχουν αρχίσει να αμφισβητούν πλέον για το μοντέλο αυτό. Δείτε τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Μέχρι ενός βαθμού αυτό θέτει εν κινδύνο και όλη αυτή την νομοθετική αρμοδιότητα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την περιφερειακή συνεργασία τόσο εντός της Ένωσης όσο και εκτός της Ένωσης. Διότι τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία είναι το αποτέλεσμα ανταγωνιστικών περιφερειακών συνεργασιών από τις δύο πλευρές, από τη μία Ρωσία, από την άλλη Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε λοιπόν ένα αρνητικό αποτέλεσμα της περιφερειακής συνεργασίας στην Ουκρανία. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ήδη και δεν ξέρουμε που θα καταλήξει αυτή η κατάσταση. Το ευρωπαϊκό λοιπόν μοντέλο, μοντέλο περιφερειακής συνεργασίας αυτή τη στιγμή αμφισβητείται και θα συνεχίσει να αμφισβητείται και στο μέλλον και από χώρε όπως η Ινδία. Επομένως έχει καταλήξει το μοντέλο αυτό είναι λιγότερο ελκυστικό από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Τώρα, για ποιο λόγο θα πρέπει να ξεκινήσουμε εκ νέου τις όλες προσπάθειες για την Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου. Όντως, η εταιρική σχέση που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση υπερβαίνει τα στενά όρια των εμπορικών ελεύθερων συναλλαγών. Δεν θα πρέπει λοιπόν να περιορίζεται μόνο από τη συμφωνία αυτή η σχέση μας. Βέβαια, θα πρέπει να δούμε και πώς έχουν τα πράγματα στην πράξη. Η βασική μας εταιρική σχέση εξακολουθεί και έχει μια έντονη οικονομική διάσταση. Και περιμέναμε ότι μέχρι το 2009, μέχρι το 2010 θα έχει ολοκληρωθεί η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών. Τελικά αυτό δεν συνέβη για διάφορους λόγους. Πιστεύω ότι αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα, τεχνικά προβλήματα και στις δύο πλευρές. Και αν αφήσουμε τα προβλήματα αυτά στους γραφειοκράτες δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε να βρούμε μια ουσιαστική λύση. Αυτό που πιστεύω το χρειαζόμαστε είναι εκ των άνω μια πολιτική όθεση. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι στην επόμενη σύνοδο κάτι ουσιαστικό μπορεί να συμβεί μπορεί να μην καταλήξουμε σε μια ευρεία συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας, αλλά και σε μια μικρότερη συμφωνία να καταλήξουμε και σε μια συμφωνία πλαίσιο απλώς να καταλήξουμε, νομίζω ότι αυτό από μόνο θα δώσει νέα όθηση στην όλη πολιτική διαδικασία. Και νομίζω ότι αυτό θα έχει ιδιαίτερη πολιτική συμβολική σημασία επίσης. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε, αυτό περιμένουμε από την Ινδία και βλέπετε ότι ο Πρωθυπουργό κύριος Ναρέντρα Μόντι ήδη έχει ανοίξει πάρα πολλούς τομείς όσον αφορά την οικονομία τώρα. Σχέσεις Ινδίας και Ρωσία. Όπως σας είπα στην ε, παρουσίασή μου αρχικά, τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία μπορεί να μην έχουν άμεση επιπτώσει στην Ινδία, αλλά εν γέννη βλέπουμε ότι η Ρωσία τελικά έρχεται όλο και πιο κοντά στην Κίνα και αυτό με τη σειρά του έχει μακροπρόθεσμα επιπτώσει στην Ινδία. Συνεπώς, απαντώ και στο τελευταίο ερώτημα το οποίο ετέθη, σχέσεις Ινδίας, Κίνας, όλα αυτά τα οποία δηλαδή απεξεργαζόμαστε στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας ή ακόμα και στα πλαίσια των χωρών BRICS. Πάρα πολλά πράγματα, όλα αυτά επηρεάζονται από την κατάσταση στην Ουκρανία. Βέβαια, η όλη ε, προσπάθεια με τα BRICS έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά καταλαβαίνετε ότι ε, η Ρωσία προσπαθεί να, χρησιμοποιεί, να χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα διαφορετικά φόρα, ιδίω όταν βλέπει ότι γίνεται μια προσπάθεια απομόνωσή τη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στην επόμενη σύνοδο. Ο Πρωθυπουργό Μόντι ε, έρχεται σε επαφές με όλες αυτές τις χώρες οι οποίες συμμετέχουν στα διεθνή αυτά φόρα. Και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ε, η Ινδία δεν περιορίζεται πλέον στις σχέσεις που έχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με κάποιους κλασικούς εταίρους της, αλλά προσπαθεί να δημιουργήσει σχέσεις και με άλλους εταίρους. Γι' αυτό το λόγο ε, είμαστε σε επαφή με τη Ρωσία, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με άλλες χώρες. Τα τελευταία δέκα χρόνια ουδέποτε είχαμε τόσο θετικές σχέσεις με όλους αυτούς σημαντικούς εταίρους ταυτόχρονα. Και επανέρχομαι έτσι στην ερώτησή σας για τις σχέσεις Ινδίας και Πακιστάν. Ξέρετε ότι υπάρχει μια τεράστια ιστορία, πάντα είχαμε καλύτερες και χειρότερες στιγμές όσον αφορά τις σχέσεις μας με το Πακιστάν, αλλά εν γέννη μπορούμε να πούμε και ήδη έχω αφιερώσει πάρα πολλές μελέτες για το Πακιστάν και έχω περάσει χρόνια και στο Αφγανιστάν. Θεωρώ ότι ε, αν αρχίσουμε και διερευνούμε λίγο περισσότερο τις σχέσεις με τις δύο αυτές χώρες, θα δούμε ότι υπάρχουν ακόμα τεράστιες δυνατότητες και ευκαιρίες που θα μπορούσαμε να, χρησιμοποιήσουμε και να εκμεταλλευτούμε. Αυτή τη στιγμή ήταν κλειστά τα σύνορα μεταξύ Ινδίας, Κίνας, Ινδίας και άλλων χωρών. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του εμπορίου περνούσε αναγκαστικά από τη θάλασσα. Ή πάρα πολλές εμπορικές συναλλαγές δεν κατέληγαν τελικά στην Ινδία αλλά σε άλλες χώρες και αναφερόμαστε σε ποσά τα οποία φτάνουν πολλές φορές ακόμα και τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν λοιπόν τεράστιες ευκαιρίες οι οποίες θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν καταφέρναμε να εκμεταλλευτούμε τις εμπορικές, οικονομικές αυτές ευκαιρίες διότι υπήρχαν πάντα πολιτικά προβλήματα τα οποία δεν μας άφηναν το κάνουμε αυτό. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι η πολιτική ηγεσία όχι μόνο στην Ινδία αλλά και στις υπόλοιπες χώρες οφείλει να συντοπίσει ότι υπάρχουν τεράστιες οικονομικές ευκαιρίες που οφείλουν και αυτοί να αξιοποιήσουν αν ε, προσεγγίσουν λίγο περισσότερο την Ινδία. Πιστεύω πάντως ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν, ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις Ινδίας-Πακιστάν. Τώρα όσον αφορά τις σχέσεις με την Κίνα. βλέπουμε ότι ε, η αρχιτεκτονική οικονομική ασφάλεια, η οποία αναδύεται σιγά σιγά στην ε, Ασία είναι διαφορετική από το μοντέλο το οποίο βέβαια ήδη υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ασία η όλη διαδικασία αυτή τη στιγμή βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Η ε, οικονομική αυτή η αρχιτεκτονική και αρτεκτονική ασφάλεια αυτή τη στιγμή δημιουργείται και χώρες όπως η Κίνα ή η Ιαπωνία θέλουν να δραματίσουν ένα τεράστιο ρόλο, συνεργαζόμενες βέβαια με την Ινδία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εταίροι, σημαντικοί παράγοντες που όλοι θέλουν να μπορούν να δραματίσουν σημαντικό ρόλο στην περιφέρεια αυτή. Η Ινδία πάντως πιστεύει ότι ε, μπορεί και αυτή να δραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Και αυτό ακριβώς φάνηκε και με την επίσκεψη του Πρόεδρου Ομπάμα στη χώρα μου. Οι Ηνωμένε Πολιτείε συνεργάζονται με την Ινδία, συνεργάζονται με την Αίζια, θέλουν να προωθήσουν περισσότερο την περιφερειακή οικονομική συνεργασία στην Ασία. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποκαθοριστεί, δεν έχει οριοθετηθεί ο ρόλος που θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένα σε αυτή την αρχιτεκτονική οικονομίας και ασφάλειας η οποία αναδύεται αυτή τη στιγμή στην Ασία. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν σημαντικές εταιρικέ σχέσεις με χώρες της Ασίας. Αλλά ποιος είναι ο στρατηγικός ρόλος που καλούνται αυτή τη στιγμή να διδραματίσουν στην περιοχή. Αυτό ακόμα δεν είναι σαφές. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ακόμα ένα πολύ σημαντικό ουσιαστικό ρόλο ή δεν αναγνωρίζεται ο σημαντικός παράγοντας σε πάρα πολλές σχέσεις που δημιουργούνται αυτή τη στιγμή με χώρες της Ασίας. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς το λόγο από την αντιπροσωπεία. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σαστέβα. Α, παρακαλώ, συγγνώμη, δεν σας είδα. Ο κύριος Επιτίδιος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον εκλεκτό ομιλητή μας ε, ποιες είναι οι σχέσεις της Ινδίας με την Ιταλία και πώς έχουν επηρεαστεί αυτές από την ε, ε, περίπτωση των ε, τριών ναυτικών. Έχει επιληθεί αυτό το πρόβλημα ή όχι και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό στη σχέση των δύο χωρών. Ευχαριστώ. χωρίς μικρόφωνο. Ε, ιδιαίτερα για αυτό το θέμα με τους Ιταλούς ε, πεζοναύτες ήταν πάρα πολύ ατυχές αυτό το γεγονός ε, στις σχέσεις Ινδίας-Ιταλίας και οι δύο χώρες κανονικά είχαν πάρα πολύ καλές σχέσεις αγαστές. Τώρα ως απόρρια αυτού του γεγονότος προσωπικά πιστεύω ότι δεν ήταν πολύ προσεκτικοί οι χειρισμοί εκατέρωθεν. Και οι Ιταλοί και οι Ινδία δεν το χειρίστηκαν καλά. Κάπως ε, πολιτικοποιήθηκε αυτό στην Ινδία το θέμα. Ιδιαίτερα το PGP όταν ήταν στην αντιπολίτευση ε, ε, είπαν ότι η κυρία Σόνια Γκάντι έχει σχέση με τους Ιταλούς και το πολιτικοποίησαν και αντίστοιχα οι Ιταλοί. Και Έγινε μεγάλη ταραχή, είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα και για τις δύο κυβερνήσεις. Ε, θα πρέπει κάπως τώρα να πέσουν οι τόνοι, οι πολιτικοί. Διαβάζει κανείς στον ειδικό τύπο ότι η ειδική κυβέρνηση ε, το έθετε ο, ο, ο Μόντι όταν ήταν στην αντιπολίτευση, το έβαζε στις προεκλογικές ομιλίες. Όταν έγινε πρωθυπουργός θέλησε να το λύσει. Αλλά και πάλι αυτό το θέμα και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεσολάβησε και άλλες εξελίξεις και αναζωπυρώθηκε και στο νότατο Ινδικό Δικαστήριο ε, όπου ασχολούνται με αυτό το θέμα. Ο, ο ένας πεζοναύτης είναι ήδη στην Ιταλία και ο άλλος είναι στην Ινδική Πρεσβεία στο Νέο Δελχή. Και αυτό είναι ένα θέμα που θα το λύσει το δικαστήριο, αλλά δυστυχώς κάπως άρχισε να επηρεάζει γενικότερα τις σχέσεις της Ινδίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον και όχι μόνο Ιταλίας, που είναι πολύ ατυχές γεγονός και εξέλιξη. Πάντως εγώ ελπίζω να λυθεί αυτό και πολιτικά. Έχει αρχίσει να επηρεάζει τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να δείξουν καλή θέληση όλα τα μέρη και ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία και η Ιταλία για να λυθεί πολιτικά πλέον αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ κύριε ε, Σάχντεβα. Θα διαβάσουμε με προσοχή τη μελέτη σας. Ευχαριστούμε και τους εκπροσώπους της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την Ινδία που μας ενημέρωσαν. Θα κάνουμε τώρα πάλι ένα μικρό διάλειμμα μέχρι τις 5 και θα ακούσουμε την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με την διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΑΚ.

Buenas tardes. Καλησπέρα σας. I speak in Spanish. Vamos... Θα μιλήσω ισπανικά. Θα περάσουμε στο τελευταίο θέμα για τη σημερινή συνεδρίαση, σε συνεργασία θυμίζω, με την αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρωπαϊκής Ένωσης Λατινικής Αμερικής. Ο κύριος Λεύτερ θα μας ενημερώσει σχετικά με τη διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΕΛΑΚ. Ήταν η δεύτερη σύνοδος, 10-11 Ιουνίου συμπροίδρευαν ε, ο πρόεδρος Τούσκ και ο πρόεδρος Κορέα, πρόεδρος της ε, Δημοκρατίας του Ισημερινού, μαζί ε, προσωπούμε το 1 τρίτο των χωρών του κόσμου και έχουμε μια κρίσιμη μάζα για να βαρύνουμε στον κόσμο. Συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος από την κλιματική αλλαγή μέχρι την ατζέντα της ανάπτυξης ε, μετά το 2015 και την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών. Υπήρξαν συμφωνίες για την ε, κρίση, για την αντιμετώπιση, ε, για τη Γιούλακ και για τους υπουργούς εξωτερικών, στους οποίους ανατίθεται να δώσουν συνέχεια στη Σύνοδο Κορυφής. Φαίνεται και πάλι ότι θέλουμε μια αμοιβαία επωφελή σχέση με αμοιβαίο σεβασμό και πάντα προς όφελος των λαών μας. Κύριε Λέφλε, παρακαλώ να μας παρουσιάσετε τα βασικά συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής, να μας πείτε πώς προτίθεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει τη συνεργασία, τι αλλαγές έχουν προκύψει και ποια είναι τα επόμενα θέματα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την τιμή αυτή να σας πληροφορήσω για τη συνεδρία που μόλις έγινε πριν από μια εβδομάδα. Γενικά, είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα της διάσκεψης. Θεωρούμε ότι παρά ορισμένα προβλήματα που θα σας αναφέρω, καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους που είχαμε θέσει στους εαυτούς μας για τη διάσκεψη αυτήν και τα τρία της μέρη πολιτικό διάλογο, οικονομικούς δεσμούς και μέλλον συνεργασία. Όπως ξέρετε εγκρίθηκαν δύο δηλώσεις, μία βραχύτερη πολιτική για της ε, συνεργασίας στην επόμενη γενεά και μία δεύτερη τη λεγόμενη δήλωση των Βρυξελών που καλύπτει όλες τις πτυχές του διαλόγου και της συνεργασίας που έχουμε μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών του ΣΕΛΑΚ. Επίσης ένα ενημερωμένο και επιυξημένο σχέδιο δράσης εγκρίθηκε και προσθέθηκαν στο παλαιότερο δύο καινούργια κεφάλαια για την παιδεία και για την ασφάλεια των πολιτών. Θα ήθελα να τονίσω ότι πιστεύουμε ότι ήταν σημαντικό βήμα προς τα εμπρός αυτό. Γιατί όλοι οι παράγοντες των διαφόρων εκδηλώσεων από την κοινοβουλευτική συνέλευση μέχρι τις ε, οργανώσεις των εργοδοτών, ακαδημαϊκούς, νεολαία, όλοι μπόρεσαν να υποβάλουν κατευθείαν στους ηγέτες τα συμπεράσματα των διαφόρων προπαρασκευαστικών συζητήσεων. Μικρό αλλά σημαντικό βήμα ώστε να συζητήσουν οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι που γινόταν δυνατόν μεταξύ τους. Θα ήθελα τώρα να σας παρουσιάσω το περιεχόμενο. Διάλογος, δεσμοί και συνεργασία. Για τον πολιτικό διάλογο, από τη μία νομίζω ότι επί της ουσίας καταλήξαμε σε σαφή γλώσσα και ορολογία για σημαντικά θέματα όπως κλιματολογικές αλλαγές, το 2020 για αναπτυξιακή πρόγραμμα και τις σφαιρικές προκλήσεις της παραγωγής και λαθρεμπορίας ναρκωτικών. που θα συζητηθούν και σε απόμενες διασκέψεις. Πράγμα που δεν ήταν και προφανές γιατί οι αρχικές θέσεις ορισμένων συνέδρων ήταν πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Έπειτα. Πολύ στεναρή στήριξη και των χωρών ΣΕΛΑ και της ενωσιακής πλευράς για τις προσπάθειες να βρεθεί η ειρήνευση μεταξύ Κολομβίας, αρχών της Κολομβίας και των ανταρτών του ΦΑΡΚ. Από την ενωσιακή πλευρά εκφράστηκε επιθυμία και προθυμία να χρηματοδοτηθεί και όλας η ειρηνευτική διαδικασία εφόσον υπογραφεί μια συμφωνία. Και τρίτον, διαδικαστικά μια συμφωνία από όλους ότι κάθε δύο χρόνια να συνεδριάζουμε δεν αρκεί και ότι επομένως οι υπουργοί θα συνεδριάζουν και μεταξύ δύο τέτοιων διασκέψεων για μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του σημείου στο οποίο θα βρισκόμαστε κάθε φορά. Η επόμενη τέτοια συνεδρίαση που θα εδράζεται στην Δομινικανή Δημοκρατία προβλέφτηκε ήδη και θα γίνει και συζήτηση για τους γενικότερους στόχους και αρχές των περιφερειακών σχέσεων. Όσο για την εμβάθυνση των οικονομικών δεσμών μεταξύ των χωρών ΣΕΛΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διάσκεψη έδωσε μια σημαντική ευκαιρία να δοθεί νέα όθηση για το εμπόριο και τις επενδύσεις μεταξύ Ένωσης και χωρών Ελλά και να επαναληφθούν ορισμένες βασικές αρχές που θα το, στις οποίες θα στηρίζεται το πρόγραμμα. Δόθηκε ιδέουσα σημασία στα σταθερά δεσμευτικά ή ρυθμιστικά πλαίσια νέα στήριξη για την πολυπλευρικότητα μεταξύ των οποίων και η έγκριση κύρωση της συνθήκης ε, του, του τελευταίου γύρου της Ντόχας και της TFA. Επίσης αναγνωρίστηκε η συμβολή του εμπορίου και των επενδύσεων στην βιώσιμη ανάπτυξη στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική και η σημασία επίσης της συνεχιζόμενης κοινωνικής ευθύνης και υπευθυνότητας. Τέλος, όλοι συμφωνήσαμε ότι η πλήρης εφαρμογή των διμερών ή περιφερειακών εμπορικών συνθήκων συνεργασίας, συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ ΕΝΟΣ και λάκ θα αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λύθο για την συνεχιζόμενη κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη των χωρών της Καραϊβικής και της Λατινικής Αμερικής. Έγινε συγκεκριμένη αναφορά και για τις ε, συνεννοήσεις Ένωσης και Μερκοσούρ και όλες οι χώρες του Μερκοσούρ δεσμεύτηκαν να προχωρήσουν μαζί καθώς και να φτάσουν πριν το τέλος του έτους σε μια θέση όπου που θα επέτρεπε την ανταλλαγή προσφορών για την προώθηση των διαπραγματεύσεων. καθώς και η σύμβαση, η προσχώρηση του Εκουαδόρ στην πολύπλευρη συμφωνία και γενικά εκφράστηκε ικανοποίηση για τη συμφωνία μεταξύ Ένωσης Μεξικού και Χιλής για τον εξυγχρονισμό ενημέρωση των συμφωνιών που, υπάρχουν, που υπήρχαν ήδη. Και αποφασίσαμε να γίνει πλήρης εφαρμογή της ε, συνθήκη σύνδεσης με τη Λατινική Αμερική και ιδιαίτερα το Περού και την Κολομβία. Έπειτα, η περιφερειακή συνεργασία, πολλά σημαντικά βήματα, πολλά. Μεγάλος αριθμός προγραμμάτων συνεργασίας, ιδιαίτερα σε, σε διπεριφερειακό επίπεδο, ανακοινώθηκαν και υπογράφηκαν στη διάσκεψη αυτή, μεταξύ των οποίων αυξημένη στήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υποδομές, εξυγίανση των υδάτων κλπ. Τέτοια προγράμματα ανήλθαν σε περισσότερα από 700 εκατομμύρια σε δεσμεύσεις από την Ένωση. Επίσης ανακοινώθηκε από την Κομισιόν ε, μια νέα, ένα νέο εργαλείο η διευκόλυνση συνεργασίας που συνδυάζει την Ένωση με μερικούς από τους πιο προωθημένους και προοδευμένους εταίρους μας. Τριγωνική συνεργασία δε με τις λιγότερο ανεπτυγμένους. Μέσω της συνεργασίας ώστε να μεγιστοποιηθεί η χρήση εμπειριών και τεχνογνωσίας με τους διαθέσιμους πόρους για να υπάρχει το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. αποτέλεσμα στις χώρες που ακόμα χρειάζονται στήριξη. Στο ίδιο πνεύμα δύο μνημόνια υπογράφτηκαν με τη Χιλή και την Ουργουάη για να εφαρμοστούν αυτά τα προγράμματα συνεργασίας. Επίσης επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή των χωρών σε ΛΑΚ στο πρόγραμμα Horizon 2020 και τα ερευνητικά του για δυνατότητες συνεργασίας και σε νέους τομείς, σε νέες διαστάσεις που δεν είχαμε ακόμη εκμεταλλευτεί μέχρι τώρα. Και σαν υποστήριξη αυτών των ιδεών και των επαφών business to business και people to people ανακοινώθηκαν 25 εκατομμύρια ευρώ συμβολή της Ένωσης για να βελτιωθεί η υψηλή ταχύτητα σύνδεση με η ευρυζωνική ταχύτητα τη σύνδεση με οπτική ίνα. Από τη Βραζιλία κυρίως προς οι άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής πρώτο τέτοιο επικοινωνιακό δεσμό μεταξύ Ένωση και Λατινική Αμερική. Γι' αυτό νομίζουμε ότι είναι και αυτό σημαντικό. Και τέλο, πάλι για τη συνεργασία που συνδέεται με επιστήμη και έρευνα. Πάνω από 9.000, σχεδόν 10.000 υποτροφίες έχουν προβλεφθεί για Λατινοαμερικανούς φοιτητές ώστε να μπορέσουν να σπουδάσουν στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια και 81,5 επίσης εκατομμύρια θα κινητοποιηθούν για τη χρηματοδότηση capacity building στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική για την ανώτερη εκπαίδευση. Άλλο βήμα που θα πρέπει να διευκολύνει κανονικά αύξηση ε, του περιβάλλοντος, απελευθέρωση θεώρησης διαβατηρίων με το Περού και την Κολομβία. Μονογραφήθηκε η συμφωνία και έχουμε πέντε συμφωνίες πλέον με ε, την Δομήνικα ε, Γρεναδίνη, ε, Αγία Λουκία και Τρινιδάδ και τον Πάγκο. Πέντε χώρες της είναι αυτές και σχεδόν ε, όλες οι χώρες ΕΛΑΚ θα ε, έχουν για σύντομη διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, άρση υποχρέωση θεώρηση διαβατηρίων. Και ελπίζω και άλλες χώρες να προσθεθούν. Ε, προσταχώς στη μεγάλη ήδη αυτή ομάδα. Ε, επιτρέψτε μου εδώ να υπογραμμίσω το εξή. Τα αποτελέσματα αυτά κατέστησαν δυνατά λόγω της καλής ή μάλλον χάρη στην καλή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλα τα θεσμικά όργανα ε, σε φάση προετοιμασίας ε, και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την ισχυρή υποστήριξη που είχαμε ανέκαθεν στους προπαρασκευαστικούς διαλόγους, ε, στην κοινοβουλευτική συνέλευση Eurolat και στις συζητήσεις που έγιναν εκεί και σε διμερείς επαφές που είχαμε με πολλούς από εσάς. Και ταυτόχρονα είχαμε και ισχυρή και υψηλή υποστήριξη και μεγάλη συναντήληψη με τα κράτη-μέλη. Πράγμα που έφερε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια ισχυρή ε, θέση και να προωθήσει τα θέματα. Γιατί είχαμε προκλήσεις, ε, δεν σας κρύβω, στην ε, προετοιμασία και μάλιστα ουσιαστικές. Γιατί υπάρχει διαφορά και διάσταση απόψεων για διάφορα θέματα. Ιδιαίτερα στην πολύ μερή ατζέντα, κλιματική αλλαγή, ανάπτυξη μετά το 2015, ε, διεθνές θεματολόγιο για τα ναρκωτικά και για άλλα. Αλλά όχι μόνο γι' αυτό υπάρχουν κάποιες θεσμικές αδυναμίες ή προκλήσεις. Από την άλλη πλευρά η ΣΕΛΑΚ είναι μια νεαρή ακόμα δομή, μια νεοσύστατη οργάνωση. Δεν έχει την ε, θεσμική αυτή μορφή που έχουμε εμείς. Δεν είναι ε, δηλαδή μόνιμος ο χαρακτήρας. Ε, είναι μεταβατική και προσωρινή κάθε προεδρία και δεν έχει ούτε την αυτονομία ούτε την εντολή να αναλάβει, να προωθήσει από μόνη της τέτοιες διαπραγματεύσεις σε επίπεδο κορυφής. Οπότε καμιά φορά ήταν ε, ετεροβαρής αυτή η διαδικασία. Εμείς είχαμε μία θέση ευρωπαϊκή και απέναντί μας 33 διαφορετικές. Τέλος, Πρόεδρε. Ε, όπως σας είπα, ε, είμαστε ικανοποιημένοι από την έκβαση της Συνόδου Κορυφής επίσης μας δίδαξε πιστεύω ότι εάν θέλουμε να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε ε, τη θέση και το ρόλο μας αλλά και την επιρροή μας στον κόσμο και στην περιφέρεια εκεί της ΣΕΛΑΚ ε, Λατινικής Αμερικής και ε, Καραϊβικής θα πρέπει να σφυριλατήσουμε πολύ γερούς διμερείς δεσμούς. Το είδαμε και στο προπαρασκευαστικό στάδιο αυτό. Και είμαι ακράδαντα πεπισμένος ότι η προσωπική ε, προσήλωση της κυρίας Μαγκερίνη και η στράτευσή της ήταν εκ των ουκάνευ για να φτάσουμε σε αυτά τα αποτελέσματα. Τέλη Ιανουαρίου βρήκε το χρόνο να πάει στη ΣΕΛΑΚ, ε, στη Σύνοδο και στην αρχή Απριλίου στη Λατινική Αμερικής ε, για να συζητήσει με τους ηγέτες και να διερευνήσει διάφορα ε, ζητήματα συνεργασίας ήταν για μας πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε σε επίπεδο υπηρεσιακών παραγόντων και υπαλλήλων να δώσουμε συνέχεια σε όλα αυτά. Θα πρέπει να το συνεχίσουμε διότι έχουν ε, δημιουργηθεί και προσδοκίες από τους εταίρους μας ε, των χωρών σε που δεν θέλουμε να απογοητεύσουμε. Θέλουμε να συνεχίσουμε λοιπόν αυτή τη συνεργασία διότι Υπάρχουν ε, και νέοι παράγοντε new kids on the block, ε, που έχουν βρει νέο ενδιαφέρον. Ξαφνικά η Κίνα ε, ανακάλυψε ότι θέλει έχει ένα φόρουμ υψηλού επίπεδου με την ΣΕΛΑΚ. Και αφού τα ξανάφτιαξε η Ουάσιγκτον με την Αβάνα, ε, έχουν επανέλθει και πολύ δραστήρια οι Ηνωμένε Πολιτείε. Υπάρχει η Ρωσία, η Ινδία και η Νότια Κορέα που ε, κάνουν ουρά για να βοηθήσουν ή για να συμμετέχουν. Δεν θα πρέπει λοιπόν εμείς να θεωρούμε τη σχέση μας δεδομένη. Θα πρέπει να την αναζωογονούμε κάθε φορά και να την εδραιώνουμε για να μπορέσουμε να έχουμε μια πολυεπίπεδη προσέγγιση και να προχωρήσουμε ε, με διάφορες υποπεριφέρειες εντός της ΕΛΑΚ και της Λατινικής Αμερικής, Κεντρικής Αμερικής και της Καραβικής. Έτσι θα μπορέσουμε να ε, συνεργαστούμε καλύτερα πολυμερώς σε διαφορά από τα θέματα αυτά. Και εκεί ακριβώς επειδή έχουμε κοινά συμφέροντα, είτε αυτή είναι η καταπολέμηση των ναρκωτικών και διακύσεις ανθρώπων ή κλιματικές αλλαγές και στα τέλη του έτους έχουμε τη σύνοδο, είτε άλλα θέματα. Έχουμε και συμφέρον, αλλά και, πώς να το πω, τη δυνατότητα να προωθήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Τώρα θα δούμε πώς θα γίνει αυτό συγκεκριμένα σε διαπεριφερειακό επίπεδο μέσω της Προεδρίας, που είναι τώρα προεδρεύει ο σημερινός, αλλά θα ακολουθήσει η Δομινικανή Δημοκρατία. Έχουμε λοιπόν μικρές εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου. Ε, η μία είναι με τις χώρες ΙΚΑ της Κεντρικής Αμερικής και η δεύτερη είναι Καριφόρουμ, είναι οι χώρες Καραϊβικής Set Και αυτά ε, θα μας ε, χαράξουν την πορεία για να δούμε πώς θα συνεργαστούμε με αυτές τις δύο υποπεριφέρειες. Έχουμε κοινή στρατηγική και κάποια συμπληρωματικά στοιχεία για την ασφάλεια των πολιτών. για θέματα εμπορίου, ανάπτυξης και άλλα. Ήδη από τώρα προετοιμάζουμε την εσωτερική εργασία μας στην Ένωση για να αναβαθμίσουμε τις συμφωνίες με το Μεξικό και τη Χιλή και για να εξασφαλίσουμε τα επόμενα βήματα με το Μερκοσούρ που θα έχουν την ίδια επιτυχία ελπίζω και πιστεύω με αυτή που φάνηκε. Αμέσως μετά τη Σύνοδο άρχισε νέος γύρος διαπραγματεύσεων για την πολιτικό διάλογο και συμφωνία σύνδεσης με την Με την Κούβα. Και ελπίζω να ε, προχωρήσουμε ουσιαστικά ε, τους επόμενους μήνες και να ολοκληρώσουμε νωρίς αυτή τη συμφωνία πλαίσιο. Και να ολοκληρωθεί αυτό το, το δίκτυο συμφωνιών που έχουμε με την περιφέρεια ΣΕΛΑΚ. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές, πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο με τους εταίρους μας από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική για να σκεφτούμε ποια θα είναι η δομή ε, και ο τρόπος συνεργασίας και αυτά θα τα συζητήσουν σε υπουργικό επίπεδο Υπουργοί Εξωτερικών το 2016 ως ένα πρώτο βήμα για την επόμενη Σύνοδο Κορυφής του 2017. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λέφτερ. Αρχίζει η συζήτηση. Καταρχάς θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ραμόν Χάουρεγγι, που είναι πρόεδρος της ε, Ευρωπαϊκής Διάστασης της Eurolat, του σκέλους αυτού. Ευχαριστώ. Κύριε Λέφλερ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω σας και την κυρία Μογκερίνη, διότι τώρα πραγματικά μπαίνουμε σε μια νέα φάση των σχέσεών μας με τη Λατινική Αμερική. Θέλω να το πιστεύω αυτό. Ήταν κακό το προηγούμενο. Τα τελευταία χρόνια δεν είχαν γίνει σπουδαία πράγματα από ευρωπαϊκή πλευρά στη Λατινική Αμερική και έχω επίγνωση της δυσκολίας που έχει ε, η κατάσταση. Το να έχει συνομιλητή μια οργάνωση που δεν είναι αρκετά οργανωμένη. Και ε, αυτό είναι πλεονασμός και είναι ασθενής. Το καταλαβαίνω αυτό και το υφίσταμαι και εγώ στη Eurolat, στις σχέσεις μας ε, με τη Λατινική Αμερική. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. ξέρω ότι είναι σύνοδος κορυφής, ξέρω πόσο κοστίζει ε, ε, να ε, πάνε όλα καλά, να υπάρχει ισχυρή παρουσία, να κοινοθέντα, ψηφίσματα, σχέδια δράσης και τα συμπαραματούντα. Νομίζω γενικά πήγε καλά η σύνοδος κορυφής και σας συγχαίρω. Και μπράβο σας που συμμετείχε και η κοινωνία. Ε, είχαμε την ευκαιρία όχι μόνο τα στελέχη και οι κυβερνήσει. Είχα εγώ τα τρία λεπτά της προσωπικής μου δόξας, μόνο ένα τρίλεπτο, αλλά εκπροσώπησα όλους τους βουλευτές της Eurolat και είπα ακριβώς και τι κάνουμε εμείς και τι κάναμε στο παρελθόν. Σας ευχαριστώ για όλα αυτά και συγχαρητήρια. Τέσσερις μικρές ερωτησούλες, τίποτα ε, και ένα σχόλιο μόνο. Μικρές ερωτησάρες. Πολύ σωστά είπατε ότι θα πρέπει να δοθεί τώρα συνέχεια στη δουλειά αυτή. Ανησυχώ και αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Θα υπάρξουν ανταλλαγές φέτος ε, προσφορών με τη Μερκοσούρ. φέτος, ναι. διότι ένα από τα σημαντικότερα ήταν αυτά ότι δεν δεσμευτήκαμε μεν, αλλά μετά τις εκλογές στην Αργεντινή μπορεί ενδεχομένως η Μερκοσούρ να μπει σε μια φάση διαλόγου επιτέλους με την Ευρώπη. Ερωτώ, μικρή ερώτηση. Θα υπάρξει ανταλλαγή προσφορών. Δεύτερη ανησυχία μου, ο Ισημερινός. Εκεί υπάρχει μια δυστοκία για τη συμφωνία με τον Ισημερινό. Εγώ νόμιζα ε, ότι αν θα έμπαινε στη συμφωνία με το Περού και την Κολομβία θα ήταν εύκολη η υπόθεση, αλλά βλέπω διάφορα προβλήματα εκεί τύπου δασμών, ε, με τον ΠΟΕ ενδεχομένω, με άλλες χώρες τις οποίες προσχωρεί. Και εγώ ανησυχώ γιατί χρειάζεται υποστήριξη ε, ο σημερινό. Το λέω ειλικρινά. Επίση ανησυχώ για τη συνεργασία με την Κεντρική Αμερική. Η Κεντρική Αμερική χρειάζεται συνεργασία πιο προηγμένη από πλευρά μα και πιο ενισχυμένη. Γι' αυτό το πρόγραμμα δράση επίση είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δοθεί συνέχεια λοιπόν στη Σύνοδο Κορυφή κύριε Λέφλερ έχει μεγάλη σημασία η στρατηγική σημασία στις μεγάλες συνόδου κορυφή, τι υπερεθνικέ, να καταλάβει ότι η Λατινική Αμερική και η Ευρώπη μπορούν να συμπίπτουν στι απόψει. και ρωτώ λοιπόν τι γίνεται εν ώψη των Παρισίων και τη Νέα Υόρκη των συνόδων για του αναπτυξιακού στόχου μετά το 2015 και μια τελευταία ερώτηση για να μην μακρηγορήσω πολύ στο σημείο 20 πρέπει να σας πω απογοητεύτηκα των δηλώσεων. Είχα την ευκαιρία να σας το πω αυτό και προσωπικά στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι έχω απογοητευτεί από την παράγραφο 20 δεν είναι ε, αυτό αντικειμενικό, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, είναι μονομερές, αναφέρει τι γίνεται στη Βενεζουέλα, αλλά καθόλου δεν συμπεριλαμβάνει την ευρωπαϊκή θέση. Έχω την εντύπωση αυτή ότι είναι έτερο βαρύς αυτή η παράγραφος και με απογοήτευσε. Δεν αντανακλά σε καμία περίπτωση το αίσθημα των Ευρωπαίων και την αίσθηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το τι συμβαίνει στη Βενεζουέλα. Ξέρω ότι δεν μπορεί να διακυβευθεί μια διακήρυξη ε, τη Συνόδου για μία παράγραφο. Το κατανοώ αλίμονο. Πώς να το πω. Προφανώς και το βλέπω αυτό ότι υπάρχουν και περιορισμοί και πρέπει να πριτανεύει ρεαλισμός. Καλύτερο θα ήταν λοιπόν να μην πούμε τίποτα άμα να πούμε αυτά τα πράγματα για τη Βενεζουέλα. Δεν μπορούμε να έχουμε μια μονομερή θεώρηση. Αυτό που μας λένε από τη ΣΕΛΑΚ. Επίσης μου έλειψε αυτή η δήλωση του κυρίου Τούσκ που έπρεπε κάπως να πάρει αποστάσεις ε, για το τι φρονούν οι Ευρωπαίοι. Λοιπόν, αυτό το παράπονο έχω να σας κάνω, το είπα και νομίζω έχει σημασία κύριε Λέφλερ να μας βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δούμε αν μπορεί να μεταβεί στη Βενεζουέλα κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο. Είδαμε το θλιβερό θέαμα. Να μην μπορέσει να πάει, φτάσει στο Καράκας ένα πούλμαν με γερουσιαστές από τη Βραζιλία. 6 Δεκεμβρίου προκήρυξαν εκλογές. Στη Βενεζουέλα. Μήπω να πάμε εκεί να ε, παρατηρήσουμε τις εκλογές για να είναι πλήρως ελεύθερες και σύμφωνα με τον νόμο της χώρας και τη δημοκρατία. Καλό θα ήταν λοιπόν μία άσκηση συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτό το λαό της Βενεζουέλας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χάουρεγγι. Ο κύριος Μιγιάν Μον. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Γενικό Διευθυντή, πρώτα απ' όλα τον κύριο Λεύτερ που ήρθε ο ίδιος προσωπικά να μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη γιατί έφτασα καθυστερημένα. Πάντως χαίρομαι που σας βλέπω και που σας άκουσα. Και επίσης χαίρομαι για την ενίσχυση των ε, σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής της ΕΛΑΚ. Ε, πολύ ωραία τα είπατε και προσυπογράφω. Ε, το πλαίσιο ποιο είναι, επανήλθαν οι Ηνωμένε Πολιτείες με την εξομάλυση των σχέσεων με την Κούβα και όλο περισσότερο ε, βλέπουμε την Νότια Αμερική και την παρουσία της Κίνας. Δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένη τη σχέση μας με τη Λατινική Αμερική ούτε να την εγκαταλείψουμε στα χέρια άλλων. Με τις χώρες αυτές μας συνδέουν τόσοι δεσμοί και ορισμένες χώρες περισσότερο από κάποιες άλλες. Και εμείς οι Ισπανοί έχουμε και δεσμούς αίματος, γλώσσας, θρησκείας και πάει λέγοντας. Γενικά η Λατινική Αμερική και η Ευρώπη συμμερίζονται πολλά οράματα, το όραμα της αξιοπρέπειας ανθρώπινης και λοιπά και πολλές αξίες. Άρα αυτό θα πρέπει να φαίνεται, όπως και φαίνεται άλλωστε στη δηλική ανακοίνωση. Να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις που έχουμε. Η Λατινική Αμερική μπορεί να είναι για την Ένωση πολύ σημαντικός εταίρος σε αυτή την προσπάθεια. Χρειάζεται παγκόσμια απάντηση και στρατηγικούς εταίρους αυτή η προσπάθεια. Ό,τι είναι λοιπόν διάλογος και προσπάθεια συντονισμού με τη Λατινική Αμερική είναι ευπρόσδεκτο. Κύριε Ελεύθερον, αυτό, από όλα αυτά που άκουσα θέλω να σταθώ σε δύο το ένα, όπω γνωρίζετε, έχει δουλέψει πολύ το Κοινοβούλιο, έρση θεωρήσεων διαβατηρίων με το Περού και την Κολομβία. Ξέρετε ότι ήταν για μας ε, μέλημα στην προηγούμενη θητεία πολλών βουλευτών. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Και ότι είναι γεγονός αυτό για στη συμφωνία με τις δύο χώρες είναι πάρα πολύ ευχάριστη είδηση. Και ε, πολύ μεγάλη ικανοποίηση για πολλούς βουλευτές και εδώ παρόντες. Κάτι άλλο που μου φαίνεται σημαντικό είναι να εμβαθύνουμε τις συμφωνίες με τη Χιλή και το Μεξικό. Ξέρετε πώς έχει διαπραγματευσει TTIP με τις Ηνωμένε Πολιτείε, με τον Καναδά κλείσαμε στην ΣΕΤΑ και με το Μεξικό η συμφωνία είναι απαρχιωμένη. Επίσης θα έχουμε συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών με τη ΣΥΠΑ και τον Καναδά και το τρίτο σκέλος της ναύτα είναι το Μεξικό που δεν θα πρέπει να μείνει πίσω και να υπολείπεται. Χαίρομαι λοιπόν για αυτή την είδηση να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και με τη Μερκοσούρ παρόλο που θα έλεγα ότι είναι ένας κήπος πολύ πιο περίπλοκος και λαβύρινθος. Και ένα τελευταίο. Και ένα τελευταίο για να συνεχιστούν οι εργασίες με τη ΣΕΛΑΚ κάθε δύο χρόνια. Είναι, ένα χρόνο έχουμε ε, Σύνοδο κορυφή, Το επόμενο χρόνο έχουμε Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών. Ε, για να μην διαταράσετε αυτή η σχέση και να μην διακόπτετε. Πολύ ωραίο. Τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια ε, για τα εξαιρετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λουίς Γκράντες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ. Και εσάς κύριε Λέφνε για την παρουσία σας και για την παρουσίασή σας. Θα φροντίσω να μην επαναλάβω αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες. Ορισμένα όμως είναι αναπόφευκτο, να τα πω κι εγώ. Υπάρχει η πολιτική δήλωση και η λεγόμενη δήλωση των Βρυξελών. Είναι αρκετά πλήρης. Ούτε με απογοητεύει τίποτα, ούτε ματέωση αισθάνομαι. Υπάρχουν πολλά στοιχεία και καινοτομίε για όλη αυτή τη διαδικασία που διαρκεί 16 χρόνια. Που δεν είναι μόνο διακηρυκτικές θέσεις, ε, υπάρχει και θάρρος και γενναιότητα και τόλμη ε, να λέμε τη γνώμη μας μέχρι και να δεσμευόμαστε. Αυτά είναι πράγματα πάρα πολύ σαφή, ξεκάθαρα και ξέρουμε τι θέλουμε στη ζωή μας. Αυτή την περιφερική συμφωνία. Βέβαια, από την άλλη υπάρχουν πράγματα που μας ικανοποιούν περισσότερο και άλλα λιγότερο. Έχουμε πλήρη επίγνωση όχι από σήμερα ούτε από χτες, από προχτές. Είμαστε παλιοί εδώ, παλιές καραβάνες και ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι και σε διπλωματικό επίπεδο να μπαίνεις σε θέματα ουσίας χωρίς να θίξεις ε, ευαισθησίες. Ε. Αλλά υπάρχουν πράγματα ε, τα οποία κανείς μπορεί να αποφύγει και κάποια άλλα που είναι αναπόφευκτα. Καλό είναι που μιλούμε για τις νέες εποχές, στη σχέση με την Κούβα είχαμε την ευκαιρία σε προηγούμενη εμφάνισή σας που μας είπατε κάποια πράγματα που παραθέτω ε, γιατί μου άρεσαν πολύ καλά. Είπατε ότι θα πρέπει να πληστούμε με υπομονή, διότι η διαδικασία αυτή και μακρά θα είναι και περίπλοκη και χρειάζεται μεγάλη ευαισθησία, αλλά έχει αρχίσει αυτή η προσπάθεια. Και όλοι έχουν την αίσθηση ότι είναι ε, μη αντιστρεπτή, μη αναστρέψιμη. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει και πώς θα μπούμε στην ουσία. Εδώ όμως κανείς δεν ομιλεί για επέμβαση, ανάμειξη στα εσωτερικά της άλλης χώρας. Το αντίθετο. Ούτε η Κούβα ε, έκανε και ένα τεράστιο επίτευγμα. Ε, με παθητικό τρόπο τα δέχεται όλα αυτά γιατί την ενδιαφέρει η δράση άλλων. Δεν έχει αναλάβει καμιά τρομερή πρωτοβουλία η Κούβα. Γι' αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε de facto και αν όχι de jure ότι ε, είναι μία κατάσταση ε, δεδομένη που δεν πρόκειται να αναστραφεί και χαίρομαι γι' αυτό. Και έχει εκφράσει και τη θέση της η Ευρωπαϊκή Ένωση για νόμους που ήταν απαράδεκτοι και ποτέ δεν δεχτήκαμε από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι γεγονό ότι θα πρέπει να περιμένουμε με υπομονή. Κάτι άλλο θετικό. Και πάλι κανείς δεν μας κατηγορεί ή κατηγορούμε κανένα για την επέμβαση ή την ανάμειξη στα ιστορικά. Είναι ο διάλογος που έγινε με τρόπο υποδειγματικό στην Κολομβία τον ενευτικό διάλογο, παρόλο που στο παρελθόν να βάγισαν κάποιες απόπειρε. Είναι κοινή λογική, θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την εξαιρετική διαδικασία, γιατί και πάλι κινδυνεύει. Είναι 50 χρόνια αυτή η ιστορία που είναι πραγματικά πόλεμος. Από τη μια είναι το κράτος που είναι, έχει τη δημοκρατική νομιμότητα, είναι έλεπτες δυνάμεις και από την άλλη είναι η ΦΑΡΚ. Και δεν μπορεί κανείς να θεωρεί ότι έχουν το ίδιο ειδικό βάρος. Ούτε ο λαός της Κολομβίας θεωρεί κάτι τέτοιο. Ούτε θα πρέπει να τη γλιτώσουν και να μην τους κοστίσει τίποτα. Ε, ατιμορρησία. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Πάντως συμφώνησαν όλοι ότι υπάρχει δυνατότητα και ε, πρέπει να το συζητήσουμε και να δώσουμε ε, υποστήριξη διαπεριφερειακή, πολιτική. Συμφωνώ με τον κύριο Χάουρεγγι διότι έχουμε ζήσει και οι δυο στη Eurolat. Εκείνο είναι πρόεδρο και εγώ είμαι κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΕΛΚ στη ναι. Eurolat. Γιατί λοιπόν έχουμε τρακ να μιλάμε για τη Βενεζουέλα. Ε, δεν είναι στην ημερήσια διάταξη. Δεν το έχουμε καταλάβει ότι συμβαίνουν πράγματα εκεί πέρα χαρακτήριστα, αχαρακτήριστα. Δηλαδή τι να λέμε ότι δεν τρέχει τίποτα. Αυτό είναι μία ψηφία του Κοινοβουλίου. Η πλειονότητα και συντριπτική μάλιστα έχει πει ότι συμβαίνουν πράγματα πάρα πολύ σοβαρά. Τώρα διπλωματικά αυτό το σημείο 20 έχει τη διατύπωση που έχει, εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε, πάντως μας απογοητεύει όντω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είναι πραγματικά κοροϊδί αυτό. Ε, είναι μπεγμός, πώς να το πω. Ε, είναι κοροϊδί εκείνος. Ε, δεν είναι δυνατό να έχουμε τόσο ισχνή διατύπωση για να διεκπαιρεώσουμε ένα θέμα με μια τέτοια διατύπωση με τόσο περίπλοκη για να μην καταλάβει κανείς τίποτα. Είναι πραγματικά απογοητευτικό. Το είπε και ο κύριος Χάορεγγι, έχει δίκιο. Εμείς ζητήσαμε διάφορα πράγματα και ευτυχώς χτες ε, ε, εξήγηλαν εκλογές 6 Δεκεμβρίου και είναι χώρος ελευθερίας επιτέλους. Εγώ δεν αρνούμε στο Μαδούρο τη δημοκρατική νομιμότητα. Ε, ε, αφισβητώ την καθημερινή διακυβέρνηση. Δεν, λέω ότι είναι αθέμητα στην εξουσία. Αλλά μικρή σχέση έχει η διακυβέρνησή του με αυτό που θεωρεί ε, φυσιολογική δημοκρατική συμπεριφορά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, επιθυμώ ειλικρινά να λυθεί δημοκρατικά το θέμα αυτό με εκλογές. Δεν χωρά καμιά αμφιβολία. Ε, πάντως, ε, ξέρω, ε, υπάρχει ματέωση και απογοήτευση για το σημείο 20. Κατά τα άλλα, τα θέματα τα είπαμε με ένα νέο στοιχείο που δεν είχαμε στο παρελθόν και τώρα σε ε, κάθε σύγχρονη κοινωνία βλέπουμε την οικολογία που χωρίς καμία αφιβολία επηρεάζει πάρα πολύ τη Λατινική Αμερική. Ποια σχέση έχει το δικαίωμα στη διαχείριση των φυσικών πόρων που είναι δημόσιο αγαθό υπέρ των λαών και ε, αυτό έρχεται σε κατάφορη σύγκρουση με κάποιες μειονότητες που θεωρούν ότι εκεί ε, το κράτος δεν έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλεύεται τους φυσικούς πόρους υπέρ του λαού. Αυτό είναι ένα θέμα που κυριαρχεί μόνιμα στη Λατινική Αμερική και θα πρέπει να το δούμε. Να δούμε ποια είναι τα περιεχόμενα και οι αξίες. Ε, ορισμένα αναφέρονται, αλλά πάλι δεν μπήκαμε στην ουσία. Θα πρέπει να είχαμε υποστήριξη στα κράτη να εκμεταλλεύονται τους φυσικούς τους πόρους πλαίσια βέβαια του σεβασμού του περιβάλλοντος. Ε, ε, γίνονται κάποιες απόπειρες πάρα πολύ δειλές και άτολμες, ίσως επειδή ξέρουν ότι υπάρχει αυτή η σύγκρουση. Κατά τάρα κύριε Λέφλερ νομίζω ότι αποκριθήκατε στην εντολή σας. Βέβαια κανείς δεν μπορεί να πιστεύει ότι θα πετύχει το τέλειο. Είναι ανέφικτο κάτι τέτοιο. Αυτές οι συνεδριάσεις διαπεριφερειακές γίνονται κάθε δύο χρόνια και ελπίζω να προχωρούν όλο και περισσότερο. Διότι υπάρχει κάτι πολύ σαφές, αλλά θέλω να το πω, γιατί λίγο το βλέπουμε. Είναι πολύ σχιζοφρενής η καιρή που ζούμε από τη μια και την άλλη όχθη του Ατλαντικού και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε Ατλαντιστές με την καλή έννοια. Δεν θα πρέπει να κοιτάμε μόνο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και προς τη Λατινική Αμερική που είναι και αυτή η Ατλαντική. Τώρα που τελειώνουν οι εργασίες στη διόρυγα του ΣΟΕΣ, θα υπάρχουν νέε δυνατότητες, του Παναμά φυσικά, συγγνώμη. Ε, θα υπάρξουν νέες δυνατότητες για να υπάρχει μια καλή συμβίωση και συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ και την παρουσίασή σας επαναλαμβάνω. Είχα ζητήσει και εγώ το λόγο και θα μιλήσω κι εγώ. Όχι ως πρόεδρος, ως απλός βουλευτής τη της ΓΚΟΕ. Νοτική αριστερά και ε, πολυφωνική αριστερά. Πρώτον, με ικανοποίηση παρατηρούμε παρατηρήσαμε τη διεξαγωγή της δεύτερης διάσκεσης κορυφής, κυρίως γιατί πρόκειται για την εξομάλυνση του γεωπολιτικού αυτού χώρου στη Λατινική Αμερική που συμβάλλει στην περιφερειακή ολοκλήρωση και κατά την άποψή μας αυτό μπορεί να αποτρέψει πολέμους και σειράξεις στην Ήπειρο αυτή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εμείς διαφωνούμε εδώ στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, δεν συμφωνούμε ε, το γεγονός ότι δεν καταλαβαίνετε τη νέα πραγματικότητα. Νομίζω ότι οι μεγάλες πολιτικές ομάδες κάνουν το ίδιο λάθος που έκαναν με την Κούβα. Είπε ο κύριος Δεκράντης κάτι για ανάμειξη στα εσωτερικά. Μέχρι ε, τώρα η Κούβα δεν είχε μετακινηθεί εφόσον δεν υπήρχε ισότιμη μεταχείριση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι περίεργο τώρα ξαφνικά ε, με την Ουάσιγκτον όλοι έχουν ξεχάσει την Κούβα και τα ρίχνουν όλα στη Βενεζουέλα. Οι ίδιοι που ήταν ε, μανιώδεις ε, αντίπαλοι της Κούβας τώρα τα ρίχνουν στη Βενεζουέλα. Έχουν γίνει λυσαλέοι πολέμοι της Βενεζουέλα. Εδώ με την Κούβα πρέπει να το πούμε εμείς οι Ισπανοί ότι έχουμε σχέσεις με την Κούβα και θα πρέπει να τις σεβόμαστε. Δεν ξέρω εάν το πήρατε είδηση, ε, αλλά στα εξωτερικά ζητήματα δεν είναι ιδεολογικό το θέμα, αλλά είναι σεβασμός του διεθνούς δικαίου. Προσπαθώ να το κάνω. Καμιά φορά δεν το πετυχαίνω κιόλας. Αυτό που δεν μου άρεσε ήταν ε, η απόπειρα από πλευράς ε, του Προέδρου Ραμόν Χαορεγγί να βάλει το θέμα της Βενεζουέλας. Επανειλημμένα το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ε, στην Ονδούρα, στο Μεξικό, στην Κολομβία συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Όταν γίνονται τέτοιες δηλώσεις ε, συζητούμε με την άλλη πλευρά με ένα σεβασμό που κατά την άποψή μου στη Βενεζουέλα δεν το δείχνεται. Είναι μια νόμιμη κυβέρνηση που βγήκε από εκλογέ, ακόμα και αν δεν σα αρέσει η ιδεολογική και πολιτική τοποθέτηση. Γίνεται λόγο για πολιτικού κρατού μένους. Μα υπάρχουν ε, περιφερειακοί οργανισμοί και ο κύριος Αμπέρτο είπε, που έγινε, είπε ότι έγινε απόπειρα πραξικοπήματος. Τι θέλετε τώρα. Και είναι περίεργο να δει κανείς τι λένε οι ε, πλειοψηφικές ομάδες εδώ. Εμείς είμαστε μειοψηφία αλλά επιμένουμε ε, και οι ε, Γκουε και οι Πράσινοι και άλλοι. Δεν υπάρχουν κοινέ δηλώσεις. Το είδαμε στο Παναμά στη Eurolat. Δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν οι πρόεδροι ακριβώς γιατί έγινε μια απόπειρα να επιβληθεί ε, από την Ευρωπαϊκή ε, ε, πλειοψηφία κάτι. Και άλλος συμπρόεδρος είπε ότι δεν μπορώ να κάνω κοινή δήλωση γιατί αυτό είναι επέμβαση και ανάμειξη στα εσωτερικά της κάθε χώρας. Ένας συμπρόεδρος από την άλλη πλευρά που μιλάει για ανάμειξη στα εσωτερικά μιας χώρας Μα αν δεν ήθελα να κάνουν εκλογές, μας λέτε δεν θέλω να κάνουν εκλογές, οι οποίες έχουν ήδη εξαγγελθεί. Ε, έλεγε ο συμπρόεδρο θα πρέπει να σεβόμαστε του θεσμού. Εμεί χαιρόμαστε για αυτή τη διακήρυξη των Βρυξελών. Για ποιο λόγο, πολύ απλό είναι. Στο σημείο 20 επαναλαμβάνουμε την απόρριψη των αναγκαστικών μονομερών μέτρων με ετεροδικία που είναι ε, αντίθετα στο διεθνές δίκαιο και η άλλη πλευρά το προσυπογράφει. Και εγώ χαίρομαι. Πάλι καλά που μπήκε αυτή η παράγραφος. Αυτό που μας εκπροσώπησε δηλαδή στην Ευρωπα... της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατάλαβα ότι πρέπει να συμφωνήσουμε με την άλλη πλευρά χωρίς ανάμειξη στα εσωτερικά της χώρας γιατί περί αυτού πρόκειται και μας το λέει και η άλλη πλευρά. Τελευταίο, για να τελειώνουμε. Στο ταξίδι εμείς είπαμε όχι. Γιατί Αντί να βρούμε λύση, να αναζητήσουμε λύση, πάτε να οξύνετε εκεί και να ξύσετε πληγές. Ε, και είναι μονομερής αυτή η προσέγγιση και παραμονές εκλογών δεν γίνεται χωρίς, δεν είναι σκόπιμο, δεν είναι ευπρεπές χωρίς τη συμφωνία της κυβέρνησης και ε, χωρίς ε, το σεβασμό να πάμε εκεί πέρα να ταράξουμε τα νερά που είναι ήδη αρκετά ταραγμένα. Ευχαριστώ πολύ. Thank ευχαριστώ πολύ αξιότιμα μέλη, για τις ρωτήσεις σας, παρατηρήσεις σας. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια σημεία, προσπαθώντας να σας απαντήσω. Πρώτον, να αναφερθώ στον φίλο μου, τον κύριο Ραμόν Χάουγγι. Μην είστε μετριοπαθείς ε, για αυτή την ε, τρίλεπτη ε, παρουσία σας. Θεωρώ ότι το μήνυμα το οποίο στείλατε ήταν πάρα πολύ καλό. Χρησιμοποίησατε πάρα πολύ καλά το χρόνο σας. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ δύσκολο να διχειριστεί κανείς μια τόσο ευρία σύνοδο με τόσους πολλούς πολιτικούς ηγέτες και τόσα πολλά διαφορετικά θέματα στη μερίσια διάταξη. Ξέρετε ότι τρία λεπτά είχαν και ηγέτες, αλλά και εσείς τα χρησιμοποίησατε πολύ καλά. Ελπίζουμε μετά την υπουργική διάσκεψη που διοργάνωσε η Επίτροπος Μάλστροπ με τις χώρες του Μερκοσούρ ότι θα καταφέρουμε τελικά στο τέλος του χρόνου να έχουμε την απαραίτητη ανταλλαγή δηλώσεων και να προχωρήσουμε περισσότερο με τη δικασία Μερκοσούρα. Η Υπουργοί και η Επίτροπος σε υψηλό βαθμό επίπεδο λένε ότι πρέπει μάλλον να εξακριβώσουν ότι όντως τηρούνται όλε οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Αλλά όχι αν έχουν γίνει οι ανταλλαγέ προσφορών και δηλώσεων. Νομίζω ότι η αποφασιστικότητα είναι σαφής και από τις δύο πλευρές. Χαιρόμαστε λοιπόν που βλέπουμε ότι οι χώρες ε, της Μερκοσούρ από κοινού και εντελώ δημόσια επανέλαβαν την στράτευσή τους προκειμένου να προχωρήσει όλη η διαδικασία ως μία ενιαία διαπραγμάτευση. Εμείς έχουμε πει επανειλημμένως ότι έχουμε συγκεκριμένη εντολή προκειμένου να διαπραγματευτούμε μια συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μερκοσούρ. Και αν δεν τροποποιηθεί η εντολή αυτή από το Συμβούλιο ή από το Μερκοσούρ, αυτό πρόκειται να κάνουμε και είμαστε πεπισμένοι ότι το να καταλήξουμε σε μια συμφωνία μεταξύ των χωρών Μερκοσούρ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ διαφορετικών περιφερειών, μεταξύ διαφορετικών οργανισμών, ε, ανταποκρίνεται στα συμφέροντα όλων. Όσον αφορά τον σημερινό, όντως αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση η χώρα και αυτό το λόγο ζήτησε αδειοδότηση κάποιων ε, μέτρων διασφάλισης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Εμείς θέσαμε απλώς κάποια ερωτήματα προς τις αρχές του σημερινού, θέλοντας να γνωρίζουμε για ποιο λόγο ζητούν επέκταση των μέτρων αυτών διασφάλισης, γιατί θα προκαλέσουν προβλήματα στην Κολομβία και στο Περού χώρες οι οποίες όπως ξέρετε πρέπει να εγκρίνουν και αυτές τα αποτελέσματα διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του σημερινού. Είμαστε πάντως πεπισμένοι ότι οι αρχές του σημερινού θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου η διαδικασία αυτή να κινηθεί ομαλά και να καταφέρουν να επανενταχθούν στο πλαίσιο συνεργασίας όπως το παρελθόν. Ο πρόεδρος Κορέα είπε και κατά τη διάρκεια της Συνόδου ότι όντως η κυβέρνησή του και η χώρα του και ο ίδιος πρόκειται να κάνουν κάτι τέτοιο έχοντας κατά νου την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη όλης της περιφέρειας. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε τώρα για τη συνεργασία των χωρών της Κεντρικής Αμερικής. Ξέρετε ότι έχουμε κάποια πολύ σημαντικά προγράμματα με όλες τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής σε περιφερειακό επίσης επίπεδο και έχουμε και κάποιες σημαντικές θεσμικές αδυναμίες τις οποίες θα πρέπει να ξεπεράσουμε αλλά και πάλι μας καθησυχάζει το γεγονός ότι υπάρχει σημαντικότατη δέσμευση από τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής στο, στην ψηλόβαθμη αυτή ξεχωριστή εκδήλωση που είχαμε με τους αρχηγούς των χωρών αυτών. για να ανταποκριθώ λίγο σε αυτά που είπε ο κύριος Μιγιάν Μόνα για την άρση υποχρέωση θεωρήσεων. Προφανώς αυτό από πρακτικής πλευράς μας επιτρέπει να έχουμε πιο έντονες επαφές με τους πολίτες από διάφορες χώρες, αλλά και συμβολικά στέλνουμε ένα μήνυμα διαλλακτικότητας και ανοιχτών συνόρων. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό με τις χώρες της Καραϊβικής, με τις πέντε αυτές χώρες Καραϊβικής και ελπίζω ότι σιγά σιγά ανάλογη πρόοδο θα σημειώσουμε και με τις υπόλοιπες χώρες της Καραϊβικής και με τις λίγες ε, ε, εναπομείνασες χώρες της Λατινικής Αμερικής για τις οποίες απαιτούνται ακόμα θεωρήσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει όμως να αναλύσουμε ακόμα περισσότερο την κατάσταση όσον αφορά την κινητικότητα πολιτών από τις χώρες αυτές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και χρειαζόμαστε και περισσότερα στατιστικά δεδομένα όσον αφορά την παράνομη είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή την παράνομη διανομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, γενικότερα, τα στατιστικά δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής δείχνουν τα πράγματα εξελίσσονται θετικά για όλες τις χώρες περιφέρειας, άρα είμαστε αρκετά αισιόδοξοι για το μέλλον και συμφωνώ απόλυτα με τις παρατηρήσεις που γίνανε για το ότι θα πρέπει να αναβαθμίσουμε τη συμφωνία που έχουμε με το Μεξικό και τη Χιλή. Πρόκειται για τις ε, πρώτες ε, πλήρης συμφωνίες σύνδεσης που είχαμε με έναν πολύ έντονο, μια πολύ έντονη εμπορική συνιστόσα οι συμφωνίε αυτέ λειτουργήσαν πολύ καλά στο παρελθόν, αλλά ήδη έχουν περάσει 15 χρόνια, 20 χρόνια από τότε που διαπραγματευθήκαμε αυτέ τι συμφωνίε. Αν δούμε πώ ήταν η Χιλή και το Μεξικό πριν από 20 χρόνια και πώ είναι σήμερα, και δείτε πώ έχει εξελιχθεί ανάλογα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Πρέπει λοιπόν να εξυγχρονίσουμε και να βαθμίσουμε τις συμφωνίες αυτές και να τις προσαρμόσουμε στη νέα πραγματικότητα των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών αυτών. Και θα πρέπει βέβαια η συμφωνία αυτή να συνάδει και με τη νέα πραγματικότητα που υπάρχει γενικότερα για τις χώρες αυτές σε περιφερειακό επίπεδο. και παράλληλα νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί και μία νέα εντολή διαπραγμάτευση για μία νέα συμφωνία με το Μεξικό και θα πρέπει να έχουμε και μία κοινή αξιολόγηση όσον αφορά τη Χιλή προκειμένου να καταλήξουμε και με τη χώρα αυτή σε μία νέα συμφωνία τα επόμενα χρόνια. Καταλαβαίνω απόλυτα τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από πάρα πολλούς για τη Βενεζουέλα. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι καταρχάς η σύνοδος αυτή ήταν διπεριφερειακή και εξέταση διπεριφερειακά ζητήματα. Αν δείτε λοιπόν τα συμπεράσματα, με την εξαίρεση της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Κολομβία και με μία μνήα που γίνεται για την έναρξη διαλόγου μεταξύ της Σαββάνας και, του, και της Ουάσιγκτον δεν υπάρχει καμία άλλη αναφορά σε διμερεί ζητήματα. Αναφέρομαι πάντα στο κείμενο των συμπερασμάτων. Είναι σαφές επίσης από πλευράς χωρών ΣΕΛΑΚ ότι ε, η επιθυμία τους ήταν να διατηρηθεί το ζήτημα αυτό σε διμερές επίπεδο και να εξεταστεί το ζήτημα αυτό ως διμερές ζήτημα, εξεταζόμενο βέβαια από μία ομάδα χωρών όπως η ΣΕΛΑΚ. Αυτό τι σημαίνει, ότι χρειάστηκε εμείς να δούμε κάποια στιγμή αν έπρεπε θα συγκεράσουμε όλες αυτές τις συγκλίνουσες ή αποκλίνουσες απόψεις ή όλες αυτές τις δεσμεύσεις ή ε, υποσχέσεις συνεργασίας, χωρίς όμως παράλληλα να εκφράζουμε κι εμείς όλες τις δικές μας ανησυχίες για κάθε ζήτημα ξεχωριστά, αφού ήταν μία εναλλακτική, ενώ η αποκλινουσες αποψεις η ολες αυτες τις δεσμευσεις η υποσχεσεις συνεργασιας χωρις ομως παραλληλα να εκφραζουμε και εμεις ήταν να μην καταλήξουμε σε κανένα τελικό και οριστικό κείμενο. Αξιολογήσαμε λοιπόν την κατάσταση και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ήταν επιθυμητό τελικά και καλύτερο να έχουμε ένα κείμενο το οποίο θα αντικατόπτριζε την γενικότερη ακόμα και διπεριφερειακή κατάσταση των σχέσεων. Αν συγκρίνετε την παράγραφο 20 για τη Βενεζουέλα με τις ε, προηγούμενες παραγράφους που έχουν να κάνουν με ανάλογες καταστάσεις όσον αφορά δηλαδή την εταιροδικία με άλλες χώρες όμως, με την Κούβα για παράδειγμα, βλέπετε εδώ πέρα ότι υπάρχουν ε, ουσιαστικές ε, διαφορές. Στις προηγούμενες παραγράφους βλέπετε ότι υπάρχει μια σύγκληση απόψεων ανάμεσα στις χώρες ΕΛΑΚ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην παράγραφο 20 η Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώνει απλώς τα όσα έχει δηλώσει η ΣΕΛΑΚ. Αλλά τα όσα λέγονται στην παράγραφο 20 εξακολουθούν και είναι απλή τοποθέτηση των χωρών ΣΕΛΑΚ και μόνο. Κατά τη διάρκεια τώρα των συζητήσεων που είχαμε, ιδίω ε, μεταξύ των ηγετών, είδαμε ότι οι ηγέτες των χωρών ΣΕΛΑΚ εκφράστηκαν με μεγαλύτερη ελευθερία και αναφέρθηκαν στις προσδοκίες, στις φιλοδοξίες, ε, τις ανησυχίες τους όσον αφορά τις διαφορετικές καταστάσεις που υφίστανται στην Ευρώπη αφενός και στη Λατινική Αμερική και την Καρυβική εφετέρου. Και όντως αυτό ακριβώς κάνα στις δηλώσεις τους. Σας, μπορώ να σας πω μάλλον ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων περιφερειακών οργανώσεων όσον αφορά την Βενεζουέλα δεν έχει τροποποιηθεί. Και αυτό έχουμε πει πάρα πολλές φορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συζήτηση που είχαμε για παράδειγμα το Μάρτιο. Και αυτό έχουμε δηλώσει πολλές φορές στο παρελθόν επίσης. Έχουμε εκφράσει μια ισχυρή ανησυχία όσον αφορά την κοινωνικονομική υποβάθμιση καθώς επίσης και την πολιτική πόλωση στη χώρα αυτή. Και έχουμε κάνει μία έκκληση για την ενίσχυση του διαλόγου ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς αποκλεισμούς. Και είπαμε επίσης ότι θα πρέπει να τηρήσουμε τόσο το Σύνταγμα όσο και την εκλογική διαδικασία στη χώρα αυτή. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς το λόγο χαιρετίζουμε το γεγονός ότι στις 6 Δεκεμβρίου θα γίνουν εκλογές στη χώρα. Θεωρούμε ότι μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί ο λαός της Βενεζουέλας να σημειώσει πρόοδο και να κινηθεί σιγά σιγά προς, ε, μία, προς ένα νεωμένο εθνικό συμβιβασμό, προς μία συνένεση, προς ένα κοινό όραμα για τη διαμόρφωση του μέλλοντός τους. Αυτό στην πράξη σημαίνει βέβαια ότι η εκλογική διαδικασία θα πρέπει να λάβει χώρα ορθά, με απόλυτη διαφάνεια. Θα πρέπει όλοι οι παράγοντες που συμμετέχουν στις εκλογές, όλοι οι ηγέτες όλων των πολιτικών κομμάτων συμπεριλαμβανομένων όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, να είναι σε θέση ελεύθερα να συνεισφέρουν στην εκλογική διαδικασία, πράγμα το οποίο δεν απόλυτα δεδομένο στις υφιστάμενες συνθήκες. Επομένως, θα πρέπει οι αρμόδιες εθνικές αρχές να εξασφαλίσουν ότι η συνταγματική εκλογική διαδικασία θα λάβει χώρα ομαλά, χωρίς προβλήματα, με απόλυτη ελευθερία και απόλυτη διαφάνεια και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί τελικά η ε, δημοκρατική διαδικασία να επικρατήσει και να δραματίσει πλήρως το ρόλο της. Εμείς πολλές φορές στο παρελθόν τονίσαμε προς τις αρχές της Βενεζουέλας καθώς και προς περιφερειακούς εταίρους της χώρας αυτής ότι είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τη διαδικασία αυτή. με τρόπο όμω που θα πρέπει να καθορίσουν οι βενεζουελικές αρχές και ε, ο λαός της Βενεζουέλας προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να εμπλακεί σε παρακολούθηση εκλογικής διαδικασίας πρέπει ουσιαστικά να κληθεί επισήμως από τις εκλογικές αρχές οποιασδήποτε χώρας. Αυτό ισχύει και ξέρετε ότι στην περίπτωση της Βενεζουέλας δεν μας έχει απευθυνθεί τέτοια πρόσκληση. Ούτε κανένας άλλος οργανισμός των ΗΕ Εθνών έχει κάνει κάτι παρόμοιο. Προσπαθούμε να δούμε αν θα μπορούσαμε εμείς με τον ένα τον άλλο τρόπο να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες περιφερειακών οργανώσεων και Απομένει να δούμε τελικά πώς θα καταφέρουμε να υποστηρίξουμε την εκλογική διαδικασία εφόσον όμως μας το ζητήσουν, εφόσον το επιθυμούν αυτό οι παράγοντες που δραστηριοποιούνται επί τόπου, στη Βενεζουέλα ή σε περιφερειακό επίπεδο. Μία τελευταία παρατήρηση όσον αφορά την Κούβα. Δεν είχαμε ξεχάσει την Κούβα στο παρελθόν, ούτε την ξεχάσαμε και τώρα. Απλώς είχαμε την κακή συνήθεια να επικεντρωνόμαστε σε κάποιες βασικές αρχές και να επεξεργαζόμαστε κάποια πράγματα μακροπρόθεσμα. Οι διαπραγματεύσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή με την Κούβα ξεκίνησαν πριν από πέντε χρόνια. Τότε αρχίσαμε να τους προετοιμάζουμε. Χρειαστήκαμε και εμείς χρόνο, χρειάστηκε χρόνο όμως και η Κούβα. Προχωράμε όμω τώρα, έχουμε τους αρχικούς μας στόχους και προσπαθούμε να δούμε πώς θα καταφέρουμε να ενθαρρύνουμε και να συνοδεύσουμε οποιαδήποτε προσπάθεια εξυγχρονισμού και μεταρρυθμίσεων στην Κούβα. Αναφέρομαι σε πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες πρέπει να λάβουν χώρα προς όφελος του ίδιου του λαού της Κούβας. Αυτός είναι ο στόχος μας, σίγουρα δεν θα επιτευχθεί εύκολα, δεν μπορεί να επιτευχθεί εν μία νυχτή, αλλά νομίζω ότι προς τα εκεί θα πρέπει να κινηθούμε στα πλαίσια της διαδικασίας που ξεκίνησε και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές ευκαιρίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να προωθήσει κάποιες θεμελιώδεις αξίες οι οποίες θα πρέπει να διέπουν και τη σχέση που έχουμε με την Κούβα καθότι η Κούβα είναι ένας πολύ σημαντικός μας εταίρος στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λέφνερ και για τις απαντήσεις που δώσατε. Θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ ε, τον ε, συμπρόεδρο τον κύριο Χάουρεγγι, να χαιρετήσω την παρουσία του. Ε, το θέμα είναι πολύ περίπλοκο. Λοιπόν, διακόπτε τη συνεδρίαση, τέλος συνεδρίασης. Επόμενη θα είναι στις 29 Ιουνίου 2015. Ευχαριστώ τους και τις Δερμηνείς και μας ευχαριστούμε.